Συνάδελφοι και συναδελφέ, παρακαλώ να αρχίσουμε. Ενώ όσο κάθεται ο κόσμος, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αλλά όμως το έξι, δηλαδή η έξι της κυρίας Μπλινκεβιτσίουτε για το πρόγραμμα της για την παιδεία, την επαγγελματική κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό και εξέταση των συμβιβαστικών αυτής τροπολογιών θα αναβληθεί για, για, για, το τέλος της συνεδρίασης. Και ο κ. Καπτουμάν ζήτησε η γνωμοδότησή του να αναβληθεί για άλλη φορά επειδή δεν υπάρχουν επειδή δεν υπάρχουν επειδή λέω δεν υπάρχουν όλες οι μεταφράσεις αν κάθισαν όλοι και όλες για θα ήθελα τώρα για τις ως ανακοινώσεις να τιμήσουμε έναν υπάλληλο που είναι ο πρώην Γενικός Διευθυντής για θέματα απασχόλησης και κοινωνικά, τον προκάτοχο δηλαδή του κυρίου Ρισέλ στην Κομισιόν, τον Ροβέρτο Βερί που έφυγε στις 26 Οκτωβρίου όλη του την καριέρα την είχε κάνει στα ευρωπαϊκά όργανα και μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ αφοσιωμένος υπάλληλος της Ένωσης πριν ασχοληθεί με θέματα απασχόλησης ήταν βοηθός του Αντιπροέδρου Ξαβιέ Ορτόλη όπου είχε ασχοληθεί με οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα. Μετά όλη του σχεδόν την καριέρα ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα και την προηγούμενη θητεία ήταν Γενικός Διευθυντής για τη μονάδα φορολόγησης και δασμών και είχε κάνει όλο τον αγώνα για να λάβει για την φορολόγηση των εταιριών και την εναρμόνιση των συνδυασμένων βάσεων για τη φορολόγηση των εταιριών. Εμείς τον γνωρίσαμε ως διευθυντή, γενικό διευθυντή για θέματα απασχόλησης και ξέρω επειδή συχνά είχα μιλήσει και με τον Επίτροπο ότι η συμβολή του εξετιμά το ιδιαιτέρως και η συνολική του γνώση για θέματα απασχόλησης και το ρόλο που έπρεπε να παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε μια στιγμή όπου η Ευρώπη γνώριζε μια κατάσταση κρίσιμης ανεργίας είχε αρχίσει μαζί με τον αρμόδιο επίτροπο να αναλύουν πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το κοινωνικό ταμείο και να έχει περισσότερη ευελιξία, αυτονομία για να ανταποκρίνεται πράγματι στις ανάγκες των Ευρωπαίων. Όσοι τον γνώριζαν ήξεραν την αξιοπρέπειά του και την αντιμετώπιση της ασθενείας γιατί ήταν μεγάλος επαγγελματίας και Ευρωπαίος αυτά ήθελα να πω και εξ ονόματος μας όλων έστειλα συλληπιτήριο τηλεγράφημα στην οικογένειά του ευχαριστώ την Κομισιόν που παρευρίσκεται εδώ θα ήθελα και εκείνοι να μεταφέρουν αυτά που είπα τώρα άλλες ανακοινώσεις άλλαξε λιγάκι το χρονοδιάγραμμα γιατί έχουμε μεγάλο φόρτο εργασίας. Θα συνεδριάσουμε εκτάκτος μαζί με τις τακτικές δηλαδή στις 6 Νοεμβρίου από τις 15 έως τις 18 η ώρα. για να συζητήσουμε μεταξύ άλλων την έκθεση της Αρκάς για τη διαβούλευση με τους εργαζομένους. 13 Νοεμβρίου και άλλη έκτακτη συνεδρίαση αλλά με μορφή κοινή συνεδρίασης με την Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Απασχόληση, όπως είχαμε κάνει και στις αρχές του έτους ειδικότερα όμως με το θέμα της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα με ανταλλαγή απόψεων με την Τρόικα. Όσοι είχαν πάει την πρώτη φορά θα θυμούνται πόσο σημαντικό είναι να θέσουμε τα ερωτήματα που πρέπει. Παρακαλώ λοιπόν να έρθετε. Τρίτον, άλλη έκτακτη συνεδρίαση. 13 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, 7 με 9 το βράδυ, όπου θα συζητήσουμε τις γνωμοδοτήσεις για την έκθεση Μπάστος επί της οποίας μόλις γνωμοδότησε η Νομική Επιτροπή. Και τη γνωμοδότηση Χόιτ για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Τελείωσαν οι ανακοινώσει. Γνωρίζετε ότι υπάρχει αναμετάδοση στο Ιντερνετ. Λοιπόν, τα πρακτικά της 6ης Ιουλίου έχουν διανεμηθεί, δεν έχω λάβει κανένα σχόλιο, επομένως εγκρίνονται. Αλλά βιάστηκα γιατί πρέπει να εγκρίνουμε και τα πρακτικά ε, γιατί καθυστέρησαν αυτό, τις 30 και 31 Μαΐου και 20 και 21 Ιουνίου. Αν θυμάστε τι έγινε τότε εκεί, τότε καλά. Εγκρίνονται. Λοιπόν, τώρα Το σημείο 4. Συμβιβασμός για την έκθεση της Μαριάννας Χάρκιν για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. 238 τροπολογίες κατατέθηκαν, κατατέθηκαν και 31 συμβιβαστικές ε, πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Είχαμε αναβάλει την εξέταση αυτή λόγω των συζητήσεων που γίνονταν στην Επιτροπή Γεωργίας που τακτικά αναβάλλονταν και εκείνες. Τώρα όμως έγιναν και υπάρχει συμφωνία για την κατανομή των δικαιοδοσιών και το χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή Γεωργίας ήθελε όλα αυτά να ξανααναβληθούν για το Δεκέμβριο. Η εισηγήτριά μας όμως επέμενε λόγω της σημασίας που έχει ζήτηση αυτή στο Συμβούλιο και είπε να τοποθετηθούμε πιο νωρίς για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει να συνεχιστεί να λειτουργεί το Ταμείο σε περίοδο όπου το Συμβούλιο φαίνεται ότι διαθέτει μια μειοψηφία που είναι αντίθετη. Βέβαια το σπανδράς μου πω τίποτα άλλο, θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να μας παρουσιάσει τις 31 συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν να παρουσιάσω του συμβιβασμού, κάποια σχόλια καταρχήν για το σχέδιο τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή Γεωργία ε, για να ενημερώσω του συναδέλφου. Ε, σύμφωνα με το σχέδιο γνωμοδότηση, όσε αναφορέ ε, στου γεωργού και στη γεωργία έχουν διαγραφεί. Έτσι λοιπόν, στι συμβιβαστικέ μα τροπολογίε κάναμε το ίδιο και αναφερόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα οι γεωργοί. Να πω ότι επίση έχουμε μία μειοψηφία ανάσχεση στο Συμβούλιο, εξακολουθεί να ισχύει, δεν σημειώνουμε καμία πρόοδο στην κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο των τροπολογιών που προτείνονται, καταρχήν ευχαριστήσω όλου του σκιώδει συζητητέ. Είχαμε αρκετέ ε, συνεδριάσει ε, και πριν την ψηφοφορία στη εξονομική θα συναντηθούμε δύο φορέ ακόμη. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα θέμα που δεν έχει επιληθεί σοβαρό και αναφέρεται στην πρόταση από τους σοσιαλιστές ε, για την αναδιάρθρωση. Έχω ε, κάποιες απόψεις λάβει, αλλά όχι από όλες τις ομάδες, δεν έχω λάβει οριστικές απόψεις και ελπίζουμε ότι στο τέλος αυτής της συνεδρίασης θα είμαι σε θέση να γνωρίζω προς τα που θα κινηθώ στο θέμα αυτό. Δεν είναι πολύ μεγάλη μεγάλη τρύπα, αλλά υπάρχει αυτή η μαύρη τρύπα στη μέση της έκθεσης. Ε, τα άλλα σχόλια και θα είμαι σύντομη γιατί θα ήθελα περισσότερο να ακούσω τους συναδέλφους σχετικά με τις προτάσεις Ένα σύντομο σχόλιο λοιπόν θέλω να κάνω έχει να κάνει με το πεδίο εφαρμογή ε, του Ταμείου Προσαρμογή τη Παγκοσμιοποίηση. Έχουμε το συμβασμό μη Ξέρω ότι κάποιοι ήθελαν να, να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογή. Εδώ δεν περιλαμβάνω το θέμα τη αναδιάρθρωση, το έχω ξεχωριστό θέμα. Όμω, πέραν αυτού, πιστεύω ότι αν διαβάσετε το συμβασμό M, το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου έχει διευρυνθεί αρκετά τις τοπολογίες που έχουμε, συμπεριλαμβάνει, που έχουμε συμπεριλάβει, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μείνει αρκετά ε, στα πλαίσια που είχε θέσει η Κομισιόν και κάποια άλλα σχόλια επιπλέον στο συνδυασμό ΓΑΜΑ, ο στόχος είναι όλοι οι εργαζόμενοι να επανενταχθούν Νομίζω ότι είχαμε καλή συνεργασία στο θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τη συγχρηματοδότηση και τους συντελεστέ, αλλάξαμε την πρόταση τη Κομισιόν. Και αυτό που θα αναφέρω τώρα είναι, ζητήσαμε 70% συγγνώμη, στα κράτη-μέλη ε, έχουν πρόσβαση στο δικό τους τομείο συνοχής. Γιατί αν δούμε τις περιοχές σύγκλησης, αυτό που είδαμε είναι ε, στις περιοχές σύγκλησης ΝΑΤΣ 2 θα σημαίνει ότι θα διατίθετον ένα ποσοστό μεγαλύτερο συγχρηματοδότηση σε χώρες όπως Γαλλία, Γερμανία, Ενωμένο Βασίλειο και θεωρήσαμε ότι δεν άρμοζε κάτι τέτοιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των εισηγητών τουλάχιστον ότι θα συμπεριλάβουμε τα ουσμέσους ε, συντελεστές ε, χρηματοδότηση ε, για τις χώρες που έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Συνοχής. Τώρα για το συμβιβασμό S, για το θέμα της επιβίωσης. Εδώ τα επίπεδα των πόρων που πηγαίνουν σε επιδόματα επιβίωσης για τους εργαζομένους είναι αρκετά σημαντικά και αυτό συμβαίνει σε κράτη-μέλη που δεν φαίνεται να είναι σε οικονομική δυσκολία. Θα ήθελα λοιπόν να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι από αυτού. Επίσης, στο συνδεσμό T, και εδώ θα ήθελα τις απόψεις σας ε, για το θέμα των εξαγορών και θα ήθελα και την άποψη της Κομισιόν, φυσικά θα τοποθετηθεί η Κομισιόν, αλλά θα ήθελα να τοποθετηθεί σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που έχω προτείνει, γιατί και αυτοί συμμετέχουν. Και θα σταματήσω εδώ για να ακούσω τι έχουν να πούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι και οι υπόλοιποι συγγητές. Mm. Παρακαλώ, θέλετε το λόγο. Η κυρία Μπάουρ. Νομίζω ότι έγινε πολύ καλή δουλειά και ευχαριστώ τη Μαριάν για το σκληρή εργασία της. Όμως, εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκκρεμούν ορισμένα ζητήματα, κυρίως όσα αναφέρθηκαν ε, το θέμα της αναδιάρθρωσης, Το συζητήσαμε αρκετά νωρίτερα, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι εφικτό τώρα γιατί δεν υπάρχει σαφή σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή για το αν είναι εφικτό ή όχι. Σε ό,τι αφορά αυτά τα επιδόματα, επιβίωση του συνδυασμό S, Πολλές φορές έχουμε δει αυτά τα επιδόματα να είναι αρκετά υψηλά αλλά ουσιαστικά θα έπρεπε να αποτελεί μία προσθήκη στο εθνικό επίδομα, το επίδομα που θα δίνεται από το Ταμείο. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι θα έπρεπε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα έπρεπε να δίνεται ένα πρόσθετο επίδομα, όχι το βασικό επίδομα, αυτό που καταβάλλεται δηλαδή από το εθνικό σύστημα. Ερώτηση όμως είναι, γιατί δεν είχα χρόνο να το ελέγξω. Άκουσα ότι είπατε ότι διαγράψετε την του Γεωργού, αλλά δεν καταλαβαίνω. Γιατί στο συμβασμό G αναφέρεται η κοινή γεωργική πολιτική. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι συμβασμοί είναι εντάξει πάνω κάτω. Αλλά θέλω να γνωρίσω αν είναι δυνατόν στο συμβασμό R. Λέμε ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν χρησιμεύει ως εργαλείο για την επίλυση της κρίσης. Εκτιμώ το ότι παντού προσθέσατε τον όρο unexpected ε, crisis, αλλά δεν το κάνατε αυτό στο συμβασμό R. Θέλω λοιπόν να συζητήσω και στο συμβασμό αυτό R να βάλετε τον όρο unexpected, πρόσμενη. Αν είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Φρεντερίκ Νταρντέν και μετά Τζιν Λαμπέρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κυρία Εισηγήτρια για όλες τις συναντήσεις που οργανώσατε για να βρούμε τους συμβιβασμούς που γενικά μας βρίσκουν σύμφωνους και για τη μείωση των προθεσμιών, για τη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που αφορούν τα μέτρα του Ταμείου Προσαρμογής. Όλα αυτά τα δεχόμαστε. Υπάρχουν όμως και ορισμένα συγκεκριμένα προβλήματα. Είπατε για την ανάληψη του εργαλείου δουλειάς από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Να δοθεί δηλαδή ειδική χρηματική βοήθεια για να αναλάβουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τον τόπο και το εργαλείο παραγωγής. Έπειτα για το συμβιβασμό σίγμα που αναφέρατε και που ζητάτε να τοποθετηθούμε μου φαίνεται ότι είναι ενδιαφέρον αλλά απλώς συμπληρωματικό συμπληρωματικό άλλων μέτρων θα μπορούσε να είναι χρήσιμο σε ορισμένες περιπτώσεις και νομίζω θα είναι αρνητικό για τους εργαζόμενους να μην υπάρχει και αυτή η δυνατότητα Όσο για το κριτήριο κρίσης που συζητήθηκε και αυτό πολύ στις προπαρασκευαστικές μας συνεδριάσεις, πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την έννοια της γενικότερης κινητοποίησης κατά της κρίσης γιατί διαπιστώνουμε ότι πολλά κράτη εξών και αυτά που είναι κατά των κριτηρίων της κρίσης τα χρησιμοποιούν για να ζητήσουν χρηματοδότηση από το Ταμείο. Άρα να διατηρηθεί. Όσο για την κατάργηση της ιδιαιτερότητας ή του ιδιαίτερου χαρακτήρα των αγροτών και αγροτισών, ε, νομίζω ότι και στην Επιτροπή ΓΕΟ συζητήθηκε το θέμα και όπως είπατε και εσείς με θελήσαμε να αναλάβουμε την αναδιάρθρωση τομέα με τομέα. Πρέπει να συνεχίσουμε να το ζητάμε αυτό, γιατί αμφισβήτητα σε ευρωπαϊκό ή ενωσιακό επίπεδο βλέπουμε να δυσκολεύονται τομείς, άλλοι να αναδιορθώνονται και από τα αιτήματα διαπιστώνουμε ότι συνεχώς σε ορισμένους τομείς επικεντρώνεται το πρόβλημα. Με μια διαδικασία λοιπόν που θα μπορούσε να επιτρέψει να υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή κάποια ταχύτερη αντιμετώπιση ή ειδική τρόπη χρηματοδότησης των αναδιαρθρούμενων τομέων θα μπορούσαμε να ταχθούμε ακόμη περισσότερο στο πλευρό των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε αυτούς τους τομείς, πάλι συμπληρωματικά. Σαν συμπλήρωμα αυτών που προβλέπει ο συνάδελφός μας Αλέξανδρος Σερκάφ στην έκθεσή του, και αυτό να το ξαναδούμε. Γιατί μου φαίνεται ότι χρήσιμο είναι, όπως είναι επίσης χρήσιμο, το Ταμείο να έχει το μέγιστο δυνατό εύρος εφαρμογής. Το Συμβούλιο, ξέρω, έχει αντιρρήσεις, ορισμένες χώρες έχουν αντιρρήσεις για το Ταμείο. Πάμε όμως στη διαπραγμάτευση με μεγάλες προσδοκίες, με φιλόδοξο πρόγραμμα και ίσως έτσι να μπορέσουμε να πείσουμε και τις πιο αμφιβάλλουσες χώρες ότι είναι χρήσιμες αυτές οι προτάσεις για να συνεχιστεί η λειτουργία του Ταμείου. Η κυρία Λαμπέρ. Ευχαριστώ, και μιλάω και στον ονόματος Σκιωδού που δεν μπορεί σήμερα να παραστεί στη συνεδρίαση. Η Μάριαν Χάκιν, σαφώς και έκανε προσπάθεια για τους για να φτάσει σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία στα οποία θέλουμε ακόμα να ξαναδούμε τη διατύπωση. Παραδείγματος χάρη όσον αφορά την συμβαστική ε που βασίζεται στην τροπολογία 100. Αναφέρεται στην κατάρτιση. Δεν έχουμε ακόμα βρει μια ικανοποιητική διατύπωση. Επίσης, συμβιβαστική τροπολογία σίγμα, S. Και εδώ Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα ακούστηκαν ότι πρόκειται για μια συμπλήρωση και όχι αντικατάσταση. Παρ' όλα αυτά όσον αφορά την κατάρτιση ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα θα πρέπει εδώ να υπάρξει μια αναφορά. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει εδώ να θεωρηθεί ότι δεν είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι αντικαθιστούμε την προηγούμενη αρμοδιότητα με αυτή τη νέα πρόταση. Είναι επιπλέον. Όσον αφορά την γεωργία, ναι, συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι εδώ υπάρχει μια ίση μεταχείριση των εργαζομένων. Συμβιβαστική τροπολογία ΤΑΦ. Τι. Εδώ δεν διαφωνούμε ως προς την ουσία, ως προς την αρχή, αλλά θα θέλαμε να δούμε κάποιες από τις πτυχές αυτού του συγκεκριμένου μέτρου που προτείνεται εδώ. Γι' αυτό και θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτηση με την εισηγήτρια. Το έθιξε το θέμα αυτό. Θεωρώ πάντως ότι κατά την άποψη τη δική μας πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση και είμαστε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ποιος άλλος ζητάει το λόγο. Η Επιτροπή. Ενδεχομένως μπορείτε να μας μιλήσετε και για το σύνολο του κειμένου, αλλά και για αυτό που είπε η κυρία Μπάουερ όσον αφορά τη χρηματοδότηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Υπάρχουν διάφορες νομοθεσίες στα κράτη-μέλη. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν αυτό θα είναι κάτι επιπλέον Έχετε το λόγο η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την επεξεργασία αυτού του θέματος. Πριν να μπω στην ουσία του θέματος, όσον αφορά την μείωση της προθεσμίας για το άρθρο 8, αυτό που είπε η ε, εισηγήτρια. Δεν ξέρω ποια θα είναι τελικά η θέση της Επιτροπής, αλλά ως προς την ουσία θεωρώ ότι μπορούμε να δεχτούμε αυτή την πρόταση, γιατί καταρχήν συμβαδίζει με την ε, δική μας θέση για το θέμα αυτό. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, κάνετε μία ερώτηση. Όλες οι υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Προσαρμογής θα πρέπει να θεωρηθούν επιπλέον συμπληρωματικές από αυτές που προβλέπονται στις εθνικές νομοθεσίες. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα μέτρα στήριξης των ε, εργαζομένων, άσχετα με την συγχρηματοδότηση, άσχετα με το αν υπάρχει συγχρηματοδότηση ή όχι, όλες αυτές οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον κανονισμό είναι επιπλέον αυτών που προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία. Και πολλές φορές ένας εργαζόμενος, για να μπορέσει παραδείγματος να υποφεληθεί από μια κατάρτιση, θα πρέπει να μπορεί να εποφεληθεί από αυτές τις ε, υπηρεσίες, άρα το Ταμείο Προσαρμογής θα πρέπει εδώ να παίξει ένα συμπληρωματικό ρόλο με αυτά που προβλέπει η Εθνική Νομοθεσία. Εισηγείτε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους, κυρία Μπάουερ. Μιλήσατε για την επιβίωση. Και άλλοι συνάδελφοι έθιξαν το θέμα αυτό. Εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι το επιπλέον, αν θέλετε, ποσό που ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη ε, σαν επίδομα επιβίωσης, ουσιαστικά εδώ φτάνει τα 60 ευρώ την ώρα. Θα δούμε τι προβλέπουν 16, 16 ε, και όχι 60 ευρώ την ώρα. Και βεβαίως εδώ θα δούμε τους κοιόδης ηθηγητές ε, και ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μία αποδεκτή πρόταση. Συμφωνώ όσον αφορά το, τη συμβαστική πρόταση G. Μπορούμε να προσθέσουμε εδώ την λέξη unexpected που λείπει από αυτήν την παράγραφο. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε όσον αφορά τους τομείς ε, στους οποίους συμβαίνει αναδιάρθρωση. Αλλά, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε τώρα για τους ε, γεωργούς. Διότι αν το κάνουμε αυτό, αυτό είναι σαν να προβλέπουμε διαρθρωτικές αλλαγές που προκύπτουν από εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό και εξαιρείται αυτός ο τομέας προς το παρόν. Θα πρέπει όμως να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν κάποιες κοινέ και αποδεκτές προτάσεις. Συζητήσαμε με την Επιτροπή για το θέμα αυτό. Όπως ξέρετε, αρχικά υπήρχε αυτός ο τομέας στην πρόταση της Επιτροπής, το πρώτο σχέδιο. Θα δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση γι' αυτό. Κυρία Λάμπερτ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε. Όντως, ε, για το θέμα της επιβίωσης, ο εργοδότης είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει αλλά θα δούμε, θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Αυτό που θέλω πάντως να πω είναι ότι ακόμα έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε πετύχει κάποια ε, σημεία. Όσοι έχουν υποβάλει τροπολογίες όσον αφορά τον αριθμό των ε, εργαζομένων που θα οδηγήσουν ε, στο BGF ήθελα να σας πω ότι δεν έχω υποβάλει συμβιβαστική τροπολογία για αυτό το θέμα διότι εδώ θα πρέπει να δούμε το θέμα των ε, επιπτώσεων όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιοχές, τις συγκεκριμένες μικρές αγορές και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως θα χαθούν. Σας ευχαριστώ. Θα εξηγήσω τη διαφωνία μου. Είναι απλώς ότι σύγκρισαν κάποια κατόφλια όχι για να καλύψουν. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σας ε, ότι ένας μηχανισμός επιτρέπει να καλύψουμε κάποια μικρή δομή. Και αν ε, ε, είναι δυνατό να υπάρξει ε, μια επαναπρόληψη, τότε θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων. Ε, γιατί εγώ δεν ξέρω μια κοπερατίβα 150 ανθρώπων, δεν ξέρω πάρα πολλές, έτσι λοιπόν ε, ίσως ε, πρέπει να υπάρχει μείωση αυτού του καταφλιού. Ίσως ε, να το δείτε και με τους σκιώδεις εισηγητές αν υπάρχει δυνατή προσαρμογή. Διαφορετικά θα ψηφίσουμε αύριο βάσει των συμβαστικών προτάσεων που μας παρουσιάσετε. Και στις 6 Νοεμβρίου ψηφίζουμε για το κείμενο αυτό. Έτσι λοιπόν, ε, ίσως ε, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω προσαρμογών. Φτάνουμε στο σημείο 5. Και εδώ να δώσω το λόγο στον κύριο Στόμας Χέντελ για να εξετάσουμε τις συμβιβαστικές ε, τροπολογίες για τις 80 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. για την έκθεση του, για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wenn sich der Rest des Saales auch... Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να περιοριστώ σε κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Πριν από δύο εβδομάδες συζητήσαμε εδώ στην Επιτροπή για το θέμα των παραχωρήσεων και συμφωνήσαμε ότι έπρεπε με συντομία, με ακρίβεια να συμφωνήσουμε. Συναντηθήκαμε με τους σκιώδεις ε, εισηγητές, τους οποίες πραγματικά τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί όντως ε, καταφέραμε να περιοριστούμε σε οκτώ συγκεκριμένες συμβιβαστικές τροπολογίες που υποστηρίζονται από πέντε πολιτικές ομάδες. Θεωρώ ότι είναι επιτυχές το αποτέλεσμα όσον αφορά την επεξεργασία αυτών των συμβαστικών τροπολογιών. Θα κάνω μια σύντομη παρατήρηση όσον αφορά το, την ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα αύριο για τις ε, παραχωρήσεις και θα ήθελα να πω πραγματικά ότι συνάδελφοι κυρίως από τη Γερμανία έχουν ε, αμφισβητήσει και υπάρχει έντονη συζήτηση όσον αφορά την ε, σημασία, την ανάγκη αυτής της οδηγίας. Και ξέρω ότι για το θέμα της ανάθεσης συμβάσεων ε, παραχώρησης υπάρχει σίγουρα πρόβλημα όσον αφορά την πλειοψηφία, την υποστήριξη από την πλειοψηφία τίθεται και θέμα επικουρικότητας των κρατών μελών όσον αφορά τις τροπολογίες που έχουν ε, υποβληθεί και από μένα και από άλλους συναδέλφους έχουν ε, χαρακτηριστεί σαν απαράδεκτες από το Προεδρείο. Και πραγματικά θεωρώ αυτό ότι είναι κατά κάποιο τρόπο εσφαλμένο. Θεωρώ πραγματικά ότι δεν ξεπέρασα τις αρμοδιότητες μου, γνωρίζω το θέμα. Όντως ε, προσπάθησα να εκφράσω την απόψή μου με πιο ολοκληρωμένο τρόπο και όχι ε, μερικός. Και αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με αυτό τον τρόπο. Τώρα, όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες, Υπάρχουν βεβαίω βεβαίως θέματα αηφόρου ανάπτυξη. είναι σαφώ κριτήρια τα οποία πάντα τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Για κάποιες από τις προτάσεις που κάνουμε, όπως παραδείγματο χάρη ένα κατάλογο κοινωνικών ε, προϋποθέσεων και κριτηρίων. Όλα αυτά θα ψηφιστούν αύριο για δύο από τις τροπολογίες που δεν αφορούν ε, από και μόνο τις ε, παραχωρήσεις. Τροπολογία 13, αδέλφου Μάνα. Εάν εδώ η Επιτροπή θέλει να ορίσει το μισ όσον αφορά την ε, ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, θα ήταν ανάλογο ή αναλόγως λογικό μα μια οδηγία να καθοριστούν με τον ίδιο τρόπο αυτές οι συμβάσεις παραχώρησης. Εγώ πραγματικά ζητώ εδώ να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία. Πραγματικά, αν η Επιτροπή κάνει μια λογική πρόταση, θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Και θεωρώ ότι θα μπορούσε να το ξανασκεφτεί ο συνάδελφος και να αποσύρει μέχρι αύριο την τροπολογία 13. Επίσης, η τροπολογία 48 της συναδέλφου Εστρέλα. Το θέμα της καλύτερης, ε, της πιο συμφέρουσας πρότασης. Ξέρετε ότι δεν αναφερόμαστε εδώ μόνο στην καλύτερη τιμή, την πιο συμφέρουσα τιμή, αλλά την καλύτερη πρόταση, την καλύτερη προσφορά και εδώ για να μην υπάρξουν παρανοήσεις, θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται μόνο για την εξέταση της τιμής. Γιατί αν μειωθεί η προσφερόμενη υπηρεσία, η όλη προσφορά είναι λιγότερο, αν θέλετε, ποιοτική, σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μπορούμε εδώ να μιλήσουμε μόνο για ανταγωνιστικότητα βασιζόμενη αποκλειστικά και μόνο στην τιμή. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μπαίνει και το θέμα του dumping. Γι' αυτό και θα ήθελα να ξανασκεφτείτε αυτήν την τροπολογία 48. Ίσως καταφέρουμε να βρούμε ίσως μια διαφορετική διατύπωση. Το εξετάσαμε και το συζητήσαμε το θέμα αυτό. Ίσως είναι λίγο αργά, αλλά τι να σας πω. Ελπίζω να βρεθεί μια άλλη διατύπωση και για την 48. Αυτά όσον αφορά την ε, συνεργασία που είχαμε με τους κοιόντες εισηγητές, με την εξαιρετική υποστήριξη της γραμματείας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους ε, για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ ο κύριος Σέρκας και κατόπιν Τόμας Μάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο γιατί η κυρία Ιστρέλα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα, βρίσκεται στο αεροπλάνο αυτή τη στιγμή, έτσι λοιπόν εγώ θα υπερασπίσω αυτά που θα ήθελε η ίδια να πει αν ήταν παρούσα εδώ. Καταρχήν θέλω να διευκρινίσω και νομίζω ότι είναι το πλέον σημαντικό ότι οι σοσιαλιστές δεν θα ψηφίσουν ε, την ε, τροπολογία αυτή που αφορά την Κομισιόν, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε στοιχεία και θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν. Από την άλλη, η κυρία Στρέλα μου είπε ότι υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με τον εισηγητή ότι υπήρξε πνεύμα συνεννόησης ε, και ανοιχτό πνεύμα γενικά και ότι θα υποστηρίξουν οι σοσιαλιστές ε, τη γραμμή των συμβαστικών προτάσεων ε, γιατί μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε την κοινωνική διάσταση αυτών των συμβάσεων. Γιατί Υπάρχει γενική συμφωνία ότι δεν είναι ίδιε όλε οι αγορέ ούτε όλε οι συμβάσει. Και αυτέ οι συμβάσει παραχώρηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ω θεμελιώδε ε, ένα στοιχείο που δεν θα αφορά μόνο το μικρότερο κόστο, αλλά τη μεγαλύτερη αξία. Θα πρέπει εμεί να φροντίσουμε να μην γίνονται τα πράγματα με έναν ανόητο τρόπο, δηλαδή να μπλέκεται η τιμή με την αξία, δηλαδή δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η τιμή που προσφέρεται σε μια ελεύθερη αγορά. Έτσι λοιπόν, για μας τους σοσιαλιστές υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που θέλουμε να υπογραμμίσουμε. Καταρχήν ότι πρέπει να είναι διαφανείς αυτές οι συμβάσει παραχώρηση Δεύτερον, πρέπει να αφαιθεί ένα περιθώριο αυτονομίας ε, στις ε, δημόσιες αρχές κάθε κράτους μέλους για να καθορίζουν ποιες είναι σε αυτές οι υπηρεσίες και ποιες είναι οι δημόσιες υπηρεσίες ε, και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο απαιτήσεων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική ε, κάλυψη των δικαιωμάτων ε, των ανθρώπων, να μην υπάρχουν διακρίσεις ε, και Τέλος, ε, το στοιχείο της μεγαλύτερης αξίας θα πρέπει να συνδυαστεί με την ποιότητα, την αηφορία και την τιμή. Αυτά τα τρία πρέπει να έχουμε υπόψη, όχι μόνο την τιμή. Έτσι λοιπόν ε, θεωρούμε ότι είναι καλή προσπάθεια αυτή. Θα συζητήσετε αύριο και με την κυρία Στρέλη της λεπτομέρειες. Εμείς θα υπερψηφίσουμε αυτούς τους συμβιβασμούς και αναμένουμε όλοι να ψηφίσουν τις συμβαστικέ προτάσεις και όχι να κατατεθεί κάποια εκτετή τροπολογία για να διαραγεί κάποιος από τους συμβιβασμού που ουσιαστικά έχουν συνθέσει τις θέσεις της πλειοψηφίας των ομάδων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμασμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τόμας, έχω μια ερώτηση. Ακούσαμε τον κύριο Σάρκας, ο οποίος εκφράστηκε υπέρ των προτάσεων αυτών των συμβιβαστικών. Θα ήθελα να ξέρω, θα πρέπει να αποσυρθεί ναι ή όχι αυτή η πρόταση αναρωτιέμαι αν θα πρέπει είτε να αποσυρθεί είτε να πούμε στην Επιτροπή ότι μπορούμε ενδεχομένως κάποια από τα σημεία στην πρόταση της Επιτροπής να τα χρησιμοποιήσουμε και με ξεκάθαρο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σημεία για να εκφράσουμε την άποψή μας. Εμείς σαν Επιτροπή Απασχόλησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κείμενο της ε, Επιτροπής, ίσως όχι τώρα και κάτι άλλο ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό στις διάφορες περιφέρειες ε, σε τοπικό επίπεδο να λάβουμε υπόψη μας την ε, επικουρικότητα. Όμως δεν μπορούμε απλώς να το αναφέρουμε αυτό. Αυτό δεν αρκεί. Και κάπου μέσα στη συμβαστική πρόταση ευεριέχεται αυτό. Αλλά για μένα είναι ένα ουσιαστικό σημείο και δεν φαίνεται αυτό. Επίσης, όσον αφορά την πιο συμφέρουσα πρόταση, όταν λέμε πιο συμφέρουσα, σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμαστε απλώς στην πιο μειωμένη τιμή. Γιατί θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να είναι λίγο πιο ε, υψηλή η τιμή που προσφέρεται, αλλά να υπάρχουν πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Κάποιες εγγύσεις, κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν εγγύσει. Όταν μιλάμε λοιπόν πιο συμφέρουσα, δεν αναφερόμαστε σε καμία περίπτωση μόνο στην τιμή. Αναφερόμαστε στην ποιότητα, στο περιεχόμενο, στο αν είναι βιώσιμη ή όχι. Mm-hmm και τα λοιπά και τα λοιπά. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει σίγουρα ε, να συμπεριλάβουμε και άλλα σημεία. Η κυρία Εστρέλα δεν είναι εδώ, αλλά για την τροπολογία 48 συμφωνώ και εγώ θα πρέπει να ξανασυζητηθεί και να αποσαφηνηθεί το περιεχόμενο. Κύρια Πρόεδρε, έχετε δίκιο θα πρέπει εδώ να τηρήσουμε τους ε, κανόνες, γιατί εδώ υπάρχουν σαφώς πολλές τροπολογίες, οι οποίες αύριο θα πρέπει να ψηφιστούν και να υποστηριχθούν με μεγάλη πλειοψηφία. Μήπως θέλει κανείς ναι. άλλος το λόγο ή καμία άλλη. Όχι, να δώσω λόγο στην Κομισιόν, αν θέλει, αν θέλει. Να δούμε όμως και αν είναι αποδεκτά. Τα βλέπω εδώ, προσέχω. Έχω εμπιστοσύνη στη γραμματεία όπως ξέρετε εκείνοι διατυπώνουν τις προτάσεις για τον καθορισμό του καθεστώτος, αν είναι αποδεκτές οι τροπολογίες δηλαδή. Και κατανοώ την άποψη της εισηγήτριας ή του εισηγητή. Όταν τραβάμε μια, ένα ανήμα πρέπει να μην ξυλωθεί όλο το πουλόβερ λοιπόν. Σε συνεργασία με τις άλλες επιτροπές, όπως θέλω κι εγώ, πρέπει να προσέξουμε να μην υπερβούμε δικαιοδοσίες. Λοιπόν, όταν ακούγονται προτάσεις που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης της ίδιας της πρότασης, τότε η δικαιοδοσία είναι η αρμόδια της ουσίας επιτροπή. Γι' αυτό και οι πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν και του εισηγητή και άλλων και που θεωρήθηκαν μη αποδεκτές, 19 τουλάχιστον. Μήπως λοιπόν η κυρία Σκικόβκα από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΚ μπορεί να μας σχολιάσει. Ναι, ένα γενικό σχόλιο και δύο ειδικά. Πρώτον, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η οδηγία αυτή αφορά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από δημόσιες αρχές και άρα είναι αρμόδια η νομοθεσία που αφορά τις δημόσιες αγορές. Με ή χωρίς την οδηγία οι κανόνες πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Η οδηγία αυτή εξειδικεύει και αποσαφηνίζει τους κανόνες ώστε οι δημόσιες αρχές και όσοι κάνουν προσφορές να γνωρίζουν τι ισχύει. Δεν έχουμε κανένα σκοπό να γίνουν όλα αυτά εκχωρήσεις. Είναι η ελεύθερη επιλογή του κοινού. Δεν πρόκειται εδώ για ιδιωτικοποίηση περαιτέρω. Προβλέπετε εδώ ένα νέο άρθρο 1α που λέει αυτά που γνωρίζετε. Όσο για τις τροπολογίες, δύο κατηγορίες βλέπω. Η μία αφορά το ίδιο το εύρος της οδηγίας και η άλλη τα κοινωνικά καριτήρια. Για το εύρος είπα ότι ακολουθούμε την οδηγή των δημοσίων αγορών. Άρα το ίδιο ισχύει για τις δημόσιες προμήθειες. Και αυτό ισχύει και για τη, τα, στα περισσότερα κράτη. Μέλη. Οι υπηρεσίες, οι περισσότερες από αυτές, ε, για αυτές έχει αποφασίσει το δικαστήριο και για τομείς που αφορούν συγκεκριμένες τροπολογίες. Προμήθεια, ε, ύδατος, αποχέτευση κλπ. Λέγεται ρητά ότι και αυτοί οι τομείς είναι στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Άρα δεν μπορεί η Κομισιόν να φανταστεί περαιτέρω αποκλεισμούς εδώ ή Υπάρχει όμως ειδικό καθεστώς για ορισμένες κοινωνικές υπηρεσίες, εφόσον έχουν ορισμένες υπηρεσίες ιδιαιτερότητες. Τέλος, ε, τις τροπολογίες για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Επίσης, ακολουθούμε τις αποφάσεις του δικαστηρίου που έχει αποφασίσει επανειλημμένος για αυτές τις υπηρεσίες. Τέλος για τα κοινωνικά. Πρώτον η οδηγία ήδη προβλέπει τη δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια εργασίας και χωρίς να ξεχνάμε το γενικό κριτήριο μπορεί να υπάρχει εξειδίκευση. Βέβαια η οδηγία αναγνωρίζει επίσης και οποιονδήποτε άλλο κανόνα κοινωνικού χαρακτήρα ήδη συμπεριλαμβάνεται στη δευτερογενές δίκαιο και άρα οποιασδήποτε τροπολογίες που μιλούν για αυτό το θέμα πρέπει να σχετίζονται, να συνδυάζονται με αυτή την οδηγία. Υπάρχει λοιπόν χώρος για να ληφθούν υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι ήδη πολλά από αυτά τα κριτήρια συμπεριλαμβάνουν στην ισχύουσα ήδη νομοθεσία. Ο κύριος ε, Σέρκας. Μόλις με ενημέρωσαν, ε, Πρόεδρε, ότι στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, κύριοι Μαν και Χέντελ αναφέρθηκαν ε, στην τροπολογία 48 της κυρίας Αστρέλα και από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόβλημα στην γερμανική εκδοχή. Ε, πρέπει να αναφέρεται το base value στα αγγλικά που είναι ο συνδυασμός της τιμής με την ποιότητα και την αηφορία. Όμως υπάρχει πρόβλημα στη μετάφραση. Σας παρακαλώ εσείς να έχετε υπόψη σας την αγγλική εκδοχή που φαίνεται ότι είναι η σωστή. Πρόεδρος. Άρα, τα αγγλικά είναι η γλώσσα αναφορά στα κοινωνικά δικαιώματα. Να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ναι, για το τελευταίο σημείο που ακούστηκε, η αγγλική μετάφραση, αν θέλετε, της τροπολογίας 48 ε, περιέχει κάποιες διαφορές σε σχέση με το γερμανικό κείμενο. Ίσως αν βασιστούμε στο αγγλικό κείμενο δεν υπάρχουν ε, τόσο μεγάλες δυσκολίες. Γι' αυτό και εγώ είπα όσα είπα, γιατί είχα μπροστά μου το γερμανικό κείμενο. Άκουσα τον Τόμας ε, Μαν. Ναι, καταλαβαίνω. Ήθελα να πω ότι σαφώς και υπάρχουν διάφοροι συνάδελφοι από διαφορετικές πολιτικές ομάδες οι οποίοι επέμειναν όσον αφορά την γενικότερη αμφισβήτηση μιας οδηγίας ε, για τις ε, συμβάσεις παραχωρήσεων. Εντάξει, το θέμα είναι ναι ή όχι δεχόμαστε αυτή τη γενική πρόταση. Μία γενική, αν θέλετε, απόρριψη περιέχει κάποιους κινδύνους. Εγώ θεωρώ ότι είναι λογικό και έχει νόημα από πολιτικής απόψεως να ξεκαθαρίσουμε εμείς, να πάρουμε θέση εμείς για το πού πρέπει να δεχόμαστε, που πρέπει να υπάρχουν συμβάσεις παραχωρήσεων και που όχι. Και να μην αφήνουμε το δικαστήριο να παίρνει αυτή την απόφαση. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η πλειοψηφία αποφασίσει να προχωρήσουμε με αυτήν την οδηγία, αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να συμπεριληφθούν τα κριτήρια αυτά και τα σημεία αυτά που έχουν μεγάλη σημασία και βαρύτητα για μας. Γι' αυτό και οι συμβαστικές τροπολογίες εδώ είναι σημαντικό να περάσουν. Euh. Και γι' αυτό και είναι πάντα σημαντικό να φτάνουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε αύριο για το κείμενο αυτό και με αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή ΙΜΚΟ θα μπορέσει να λάβει υπόψη τη δική μας ε, ψηφοφορία το Δεκέμβριο. Και τώρα περνάμε στο σημείο 7. Όπως είπαμε το σημείο έχει συζητηθεί στο τέλος συνεδρίασης και θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Jean Lambert για τις συμβιβαστικές τροπολογίες 7 στον αριθμό. που έχουν υποβληθεί για το θέμα του προγράμματος Δικαιώματα και Ιθαγένεια για την περίοδο 2014-2020. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση. Επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η συγγήτρια είναι η συνάδελφος Κίνγκα Κόντς. Εύκολο λοιπόν να συνεργαστούμε με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η κυρία Λάμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Στην περίπτωση αυτή, η συνεργασία μεταξύ των Επιτροπών ΛΥΜΠΕ και Επιτροπής Απασχόλησης είναι καλή Είχαμε μια συνεδρίαση με του σκιώδη ε, τη Επίτροπή Λιμπέ για να δούμε τις πιθανές συμβαστικές τροπολογίε ε, που καταρτίζουν αυτοί. Όπως φαντάζεστε αυτοί έχουν πολύ περισσότερε τροπολογίε στο συνολικό φάκελο. Και ήδη σε αρκετά θέματα φαίνεται να υπάρχει συμφωνία μέσω συμβαστικών τροπολογιών ε, και ήδη λαμβάνονται υπόψη. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η καλή συνεργασία. Αυτή η νομοδότηση, μάλλον ε, αυτό το θέμα το εξετάζουν ε, τρεις επιτροπές. Γι' αυτό το λόγο, στον ε, κατάλογο ψηφοφοριών θα δείτε ότι υπάρχουν τρεις τροπολογίες, οι 42, 43 και 44 που φαίνεται να είναι απαράδεκτες και σχετάζονται με ένα εκτιμώντας. Και αυτό οφείλεται στην ε, κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιτροπών. Το θέμα λοιπόν ε, το παρακολουθούμε, απλώς παρακολουθείτε σε άλλη επιτροπή. Ήθελα να πω δύο λόγια για τον κατάλογο ψηφοφοριών ε, για την τροπολογία 46 του κυρίου Χάντελ, άρθρο 4, παράγραφος 1C, 1Γ, που σχετίζεται με ένα τμήμα του πεδίου αυτού του ταμείου. Αν ε, δούμε τα θέματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών και τα δικαιώματα των καταναλωτών, έχουν υπάρξει κάποιες συζητήσεις και σε αυτή την Επιτροπή και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και με την Κομισιόν για το αν αυτό είναι το κατάλληλο σημείο να αναφέρεται αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ότι ορισμένε από τις πτυχές που σχετίζονται με τα δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να παραμείνουν σε αυτό το φάκελο. Δεν ε, υπάρχει κατάλληλο ε, χώρο να μετακινηθούν ε, σε μπλοκ ε, όλα αυτά τα θέματα όπως σε άλλο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, στο κατάλογο ψηφιλίου νομίζω ότι από μένα ως εισηγήτρια εκείνη η μόνη ένδειξη για το τι θα πρέπει να καταψηφίσουμε. Για τα υπόλοιπα υπάρχει συμφωνία. Αλλά σας εξήγησα το λόγο. Γιατί φαίνεται ότι δεν μπορούμε να έχουμε μετακίνηση σε μπλοκ. Σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες έχουμε 7 και οι 7 ε, βρίσκουν ε, σύμφωνα 5 πολιτικές ομάδες και ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που έκαναν ε, το συντονισμό σε σχέση με τη διατύπωση στο συμβασμό Β, που σχετίζεται με το άρθρο 5 και το συμβασμό Ή που σχετίζεται με το 4-1-β. Είχαμε κάποια ζητήματα που αναφέρθηκαν. Σημεία που θέλουμε να αποσαφηνίσουμε ότι δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές οι διακρίσεις. Αυτό έχει να κάνει και με τη συνθήκη και με τη χάρτα. Έτσι λοιπόν τώρα στις τροπολογίες αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τη γνωμοδότηση της χάρτας και να λέμε such as και όχι in particular. Έτσι ώστε να ακολουθούμε την ε, υφιστάμενη νομική διατύπωση. Υπήρξε και ένα άλλο θέμα για την ε, ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων που μετακινούνται στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πάλι στο συμβασμό ΓΑΜΑ εκτιμώντας 10 και στο συμβασμό Ε για το 4.1β βρήκαμε μία διατύπωση η οποία τώρα είναι σαφής δεν ε, προσπαθεί να κάνει εικασίες για το αποτέλεσμα άλλων ε, φακέλων που εξετάζουμε στην Επιτροπή. Δηλαδή αναφερόμαστε σε διακρίσεις ε, βάσει της εθνικότητας ε, και σε τομείς που αφορούν ε, την αγορά εργασίας. Συμφωνούμε ότι πρόκειται για την αγορά εργασίας και όχι για τις υπηρεσίες. Δηλαδή δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε αυτό με το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων. Εδώ μιλάμε για τα δικαιώματα των ατόμων. Και κάτι ακόμη να πω για το συμβασμό που σχετίζεται με το εκτιμώντας 5. Ξέρω ότι δεν το κάνουμε αυτό στην Επιτροπή συνήθως. Εδώ εισάγεται ένα άλλος τομέας μη εισαγωγή διακρίσεως, όπου δεν μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία μεταξύ των ομάδων. Επομένως, είναι πιο εύκολο να το ψηφίσουμε αυτό ως ξεχωριστό ζήτημα και να δούμε τι υποστηρίζει η πλειοψηφία. Παρά να πρέπει να διαγράψουμε ένα μεγάλο βαθμό συμφωνίας που είχαμε πετύχει ήδη. και να ψηφίσουμε κάποιες τροπολογίες ε, που θα θεωρούνται χάσιμο χρόνο από ορισμένους. Έτσι λοιπόν, τροπολογία 24 που σχετίζεται με την ε, ταυτότητα των ε, φύλων αποτελεί προσθήκη. Αυτά ήθελα να πω εγώ επεξηγηματικά. Και όπως σας είπα, ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τη συνεργασία που είχαμε. Και νομίζω ότι έχουμε μία σαφή γνωμοδότηση τώρα. Και θα λάβουμε υπόψη φυσικά και τις ε, σκέψεις της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών ε, και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και φυσικά θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με το Συμβουλίο. Ευχαριστούμε πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήδη από την προηγούμενη συνεδρίαση είχα ευχαριστήσει την εισηγήτρια, την ξαναευχαριστώ και πάλι για την καλή συνεργασία και τους συμβιβασμούς ιδιαίτερα ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θέλω όμως να τονίσω το εξής. Ο συμβιβασμός ε δεν με ικανοποιεί. Μπορεί βέβαια κανείς να τον ερμηνεύσει με διάφορους τρόπους, αλλά η αρχική διατύπωση που έλεγε ότι τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα ή μάλλον θα έπρεπε να μπορούν να εγγυώνται την ισότητα, την ίση μεταχείριση είναι πολύ καλύτερη αντί αυτήν που λέει να καταργηθούν όπως λέει. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η πρώτη αρχική διατύπωση είναι σαφέστερη, ζητάει αυτό που ζητάει με τρόπο πολύ πιο ρητό. Αφού όμως είναι συμβιβασμός, εάν τον δέχονται όλοι ελπίζω να συμφωνήσουμε ότι οι εργαζόμενοι όπου και να διαβιούν ή να εργάζονται πρέπει να τη χάνουν ίσης μεταχείρισης Έχω αμφιβολίες λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά είμαι υπέρ του συμβιβασμού. Μάλιστα, Αριάν Αρκίν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντοτε πιστική η συγγήτρια, την ξέρω. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με τους συμβιβασμούς και νομίζω ότι εκφραζόμαστε αρκετά στεναρά για την ίση μεταχείριση και παραπέμπουμε και στη συνθήκη της Λισαβόνας και στη χάρτα των θεμελιωδών. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Επίσης ο συμβιβασμός γάμα με ικανοποιεί και για την τροπολογία 24 και αυτή μπορούμε να τη δεχτούμε αν και καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο διαχωρίστηκε από τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία. Μάλιστα η Κομισιόν, η κυρία Πιπίδου. Ναι, γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Μερικά γενικά μόνο σχόλια. Εδώ χρειάζονται ορισμένες ε, τεχνικές διευθετήσεις ώστε να σεβόμαστε τα όρια που θέτει η επιλεγμένη νομική βάση και επίσης για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν επικαλύψεις με άλλα προγράμματα. Ευχαριστώ. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να ξαναδώσω λόγο στην κυρία Λαβέρ. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Τους ευχαριστώ όλους και όλες για την ευελιξία τους, όσο δε για τη διευθέτηση των τεχνικών λεπτομεριών που ανέφερε η Κομισιόν. Αυτό θα γίνει από την Επιτροπή ΕΛΕΦ και από περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Από εμά την απασχόληση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δοθεί μια γενικότερη κατεύθυνση, την οποία να δεχόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο αυτή τη γνωμοδότηση. Τώρα ερχόμαστε στο σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Βερονίκ Λόπης Φοντανιέ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποθέσεων Θαλάσσης και Αλλιευτικών. Ο κύριος Αλέν Καντέκ είναι ο αρμόδιος επί της ουσίας. Όσο δε για την έκθεση ε, η γνωμοδότηση Φοντανιέ, 76 τροπολογίες κατατέθηκαν, 80, από την συγκήτρια και 84 από τους συναδέλφους και καταλήξαμε σε 12 συμβιβαστικές. Το λόγο έχει τώρα η συντάκτρια της γνωμοδότησης. Εδώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, Πιστεύω ότι έγινε προσπάθεια να καταλήξουμε σε συμφωνία. Καταρθώσαμε να καταλήξουμε συνδεσμούς με τέσσερις ομάδες. Ε, σε αυτές τις συμβεστικές προτάσεις ε, δώσαμε έμφαση στο θέμα της απασχόλησης, κυρίως ε, μιλώντας για την καταπολέμηση της φτώχειας, μιλώντας για τις ευπαθείς ομάδες εγώ νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά. Πρέπει να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες και ανεξαρτήτως αυτών των τριών τροπολογιών υπάρχουν αυτών των τριών συμβιβαστικών τροπολογιών υπάρχουν και αρκετές τροπολογίες που δεν τις αποσύραμε και αποτελούν αντικείμενο συμβιβασμού γιατί θα ψηφιστούν ως έχουν και θα υπερψηφιστούν οι περισσότερες γιατί εγώ νομίζω ότι βελτιώνουν όλο το κείμενο συνολικά. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που δεν μπορούσα να δεκτώ στις τροπολογίες, κυρίως όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίζεται να διατηρείται ο όρος αυτός και επίσης ε, για την αιρεσταχνική αλία θα πρέπει να την προστατεύσουμε γιατί είναι η αλία που δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας και επίσης ευνοεί και την απασχόληση στις ε, οικογένειες. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι συνάδελφοι θεώρησαν ότι θα έπρεπε να υποστηριχθεί τα μάλα αυτή η αεραστεχνική έλεια. Και πάλι να σας ευχαριστήσω όλους. Tak for formand, og tak til øh, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη συνεργασία μας. Κατά την άποψή μου πρέπει να προσδώσουμε μια κοινωνική διάσταση στο ταμείο αυτό. Το ταμείο αυτό πρέπει να βελτιώσει τις συνθήκες για τους εργαζομένους και θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι συμβάσεις ε, και ο κοινωνικός διάλογος. Θα πρέπει επίσης ε, να υποστηρίξουμε την ε, βελτίωση των συνθήκων εργασίας, γιατί η αλία είναι ένας δύσκολος τομέας και συχνά ενέχονται κίνδυνοι στη θάλασσα, αλλά και στην ξηρά. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ισχυρή αλία και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε και την καινοτομία στον τομέα. Επίσης, υπογραμμίσαμε ότι ήταν σκόπιμο οι κοινωνικοί εταίροι να συμπεριλαμβάνονται στο έργο αυτό. Αυτό είναι πάντοτε σημαντικό όταν μιλάμε για δύσκολες συνθήκες εργασίας. Ο συμβασμός όμως που βρήκαμε μας επέτρεψε να εξισορροπήσουμε τις διάφορες απόψεις και να έχουμε μια ισχυρή βάση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή Ελίας. Και πάλι όμως θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της και σας ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Πρόεδρος, θέλει κάποιος άλλο το λόγο? Όχι. Όλα πήγαν καλά στο φάκελο αυτό. Θα ψηφίσουμε αύριο. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης και εδώ σας πρότεινα να εξετάσουμε τις 22 συμβαστικές τροπολογίες που εκπονήσαμε με τους σκιώδεις εισηγητές για την γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΕΚΟΝ προς μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Σε μένα αναθέσατε την ευθύνη κατάρτισης της έκθεσης αυτής. Καταρχήν να ευχαριστήσω και πάλι τους σκιώδους, τους σκιώδεις εισηγητές. Είχαμε μια πολύπλοκη διαδικασία Δηλαδή στην αρχή είχαμε μια δυσκολία καθώς ε, στην Επιτροπή Εκών πρόκειται για μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας ε, που αποτελείται από δύο μέρη. Ένα τμήμα που έχει τη μορφή κλασικού ψηφίσματος όπως το γνωρίζουμε και προβαίνει στην διατύπωση συγκεκριμένων συστάσεων. Έτσι λοιπόν ε, για να συστήσουμε, να καταρτήσουμε την έκθεση με ένα τρόπο συμβατό ε, με τη διαδικασία που ακολουθήκε στην ΕΚΟΝ ε, έπρεπε να έχουμε ένα ειδικό τρόπο σύνταξη. Και η Επιτροπή ΕΚΟΝ μπορούσε να συνεισφέρει. Και η συνεισφορά αυτή θα ε, ξανατονίσει την κοινωνική πτυχή ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων ε, στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Καθώς πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία αναφορά στην κοινωνική διάσταση. Εδώ στις συμβαστικές τροπολογίες ξαναβρίσκουμε την αναφορά στη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Ξέρουμε ότι έχουμε τρεις σημαντικούς στόχους εκεί, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναφορά σε αυτό το φαύλο κύκλο και στα μετρελιτότητα και την ύφεση, βρήκαμε ένα συμβιβασμό, διευκρινίζοντα ότι πρόκειται για μια κατάσταση που οδηγεί σε φαύλο κύκλο ορισμένα κράτη-μέλη όχι απαραίτητο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Κατόπιν. Με πολλές ομάδες και με ορισμένα μέλη του ΕΛΚ συζητήσαμε αυτή την ε, κοινωνική πτυχή Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η νέα κοινωνική πτυχή της νομισματικής και οικονομικής ένωσης, δίνοντας έμφαση στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, χωρίς όμως ε, αυτό να αντικαθιστά κάθε νομοθετική πρωτοβουλία. Χωρίς δηλαδή να οδηγούμαστε σε μια τέτοια αναγνώριση που θα απαγόρευε την παρέμβαση του νομοθέτη. Και κατόπιν ε, λάβαμε και πάλι υπόψη μια πρόταση της Κομισιόν στο πλαίσιο του and Job Recovery προς ανάκτηση των θέσεων εργασίας όπου είχε προτεθεί η σύσταση μιας νέας τριμερούς δομής ε, για να υπάρχει καλύτερη διεπαφή μεταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού επίπεδου στα κοινωνικά θέματα. Δεν θα αναφέρω όλα τα στοιχεία του συμβιβασμού, αλλά αυτές οι συμβαστικές προτάσεις ε, εκπονήθηκαν ε, δίνοντας ε, έμφαση στο θέμα της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες ή στον αξιοπρεπή μισθό. Μια άλλη συμβαστική πρόταση έχει να κάνει με το θέμα της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων και να δούμε τι, πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα των αποσπασμένων εργαζομένων στην περίπτωση αυτή. Εκεί βρήκαμε μια συμβαστική λύση που μας ε, επιτρέπει να μην ε, έρθουμε σε αντίθεση με την έκθεση της κυρίας ε, Τσαπιλοπιέσκα. Αλλά να μιλάμε για μια ορθή, σωστή αμοιβή των εργαζομένων. Για να παρουσιάσω τις κυρίες συμβαστικές τροπολογίες, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του άρθρου 9 της συνθήκης. Εδώ έχουμε συμπεριλάβει κάποιες ανησυχίες της ε, κυρίας Σάια καταρχήν ε, που ευθύθηκαν και από το ΕΛΚ στη συνέχεια για το θέμα της ε, συνεισφοράς ημί του δημοσίου στη μείωση του ελλείμματος, των δημοσίων Δεπανών στη μείωση του ελλείμματος και κατόπιν αιτήματο των πρασίνων εντάξαμε μία ανησυχία για την πραγματική αξία του μισθού. Δηλαδή όχι ως προσαρμογή αλλά ως μέσο επιβίωσης των εργαζομένων. Και υπάρχει και μια σειρά συμβιβαστικών τροπολογιών που αφορά το εξή ότι θα πρέπει ε, να έχουμε καλύτερες ε, συνθήκες ε, διακυβέρνησης ό,τι αφορά του τομεί αρμοδίτητων αυτή τη επιτροπή. παράλληλα με την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, κανεί δεν θα το κάνει αντί για μας. Επίση, βρήκαμε μια συμβαστική λύση. κυρίως με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους για τη συνεισφορά του κοινωνικού μοντέλου για τη μείωση των ανισοτήτων και της ε, δημιουργίας ε, κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης έχουμε και ένα ακόμη σημαντικό συμβιβασμό που αναφέρεται στο ζήτημα των εθνικών σχεδίων για την απασχόληση. Όπως ξέρετε, αυτό το έγγραφο θα πρέπει να εκπονηθεί από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης όλα τα, δεν, τα δεν το έχουν κάνει όλα τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν ε, τελικά δεν φαίνεται να δίνει και τόση σημασία στο σεβασμό αυτής της υποχρέωσης από την πλευρά των κρατών μελών και εμείς υπενθυμίζουμε εδώ στις συμβαστικέ τροπολογίες ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο του μηχανισμού κυρίως στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το συμβασμό ΒΕ Εδώ με τους φιλελευθέρους ε, προσεγγίσαμε το θέμα του Συμφώνου Ανάπτυξης, έτσι όπως ειτήθηκε από το Συμβούλιο της 28-29 Ιουνίου, ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά θα πρέπει και να συμπληρωθεί από ένα σύμφωνο κοινωνικού χαρακτήρα. Και όλα αυτά που σας ανέφερα βρίσκονται στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης, ε, στις συστάσεις ε, δηλαδή, αυτές οι αυτές. Δεν θα τα επαναλάβω όλα, απλώς να σας πω ότι μέσω των συστάσεων αυτό παρουσιάζεται το ζήτημα ανάληψης μιας πρωτοβουλίας υπέρ των νέων, Νομίζω ότι εδώ έχουμε δύο προτάσεις αρκετά πρωτότυπες, σχετικά καινοτόμε. Σε μια συζήτηση που υποστηρίχθηκε από πολλούς συναδέλφους, η πρώτη είναι η ιδέα ότι χρειαζόμαστε, πρέπει να σκεφτούμε μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι να έχουμε μια γενική ευρωπαϊκή επιθεώρηση εργασίας, αλλά ένα φορέα συμπληρωματικό που θα μπορούσε ουσιαστικά να στηρίζει τις εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας. Και ξέρετε ότι ε, έχουμε διάφορα δικαιώματα, καθώς έχουμε και πολλούς αποσπασμένους εργαζομένους, αλλά έχουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση δυναμή της σημερινής νομοθεσίας και όλα αυτά θα έπρεπε να ελευθούν ή να μπορούν να γίνουν αντικείμενο επιθεώρησης επιτόπου. Και μια δεύτερη πρόταση για την οποία ευχαριστώ τους συναδέλφους που θεώρησαν ότι ήταν χρήσιμη να διατυπωθεί στην έκθεση αυτή είναι η εξή: ε, ότι εκεί ε, όπου έχουμε ε, την δυνατότητα της κίτρινης κάρτας δηλαδή να μπορούν τα εθνικά κοινοβούλια να ζητήσουν ε, την απόσυρση μιας πρώτης κομισιόν ε, ή ε, την τροποποίηση της πρότασης αυτής θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια πράσινη κάρτα που θα επιτρέπει στα εθνικά κοινοβούλια να απευθύνονται στην Κομισιόν και να τη ζητούν να εκπονήσει μια πρόταση, μια νομοθετική πρόταση πρωτοβουλίας γιατί όταν, ε, όταν θεωρούν, μάλλον στην περίπτωση που θεωρούν ότι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρξε αρκετά ευρύ ε, συμβιβασμό για να είμαι σίγουρη για την επιτυχία της πρότασης. Όμω, ε, έχουμε και το θέμα της αποζημίωσης του επιδόματος ανεργίας Εκεί εξελίσσονται οι συζητήσεις και ο ίδιος Επίτροπος παρακολουθεί τις τροπολογικές ε, πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον τομέα αυτό και αν εμείς από την πλευρά της δικής μας ε, Επιτροπής, ε, αν δεν το καταφέρουμε θα θεωρήσω ότι είναι κρίμα. Και πάλι ευχαριστώ όλες τις ομάδες για την κατανόησή τους, για τη μέθοδο που ακολουθήθηκε και Ζητώ συγγνώμη. Γιατί αυτή η διαδικασία ήταν δύσκολη αρχικά. Γιατί έγιναν κάποιες αλλαγές στην πορεία. Να δώσω το λόγο σε το επιθυμούν. Καταρχήν, ο κύριος Όρη και κατόπιν ο κύριος Σέρκας. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι ήμασταν εξαιρετικά χαλαροί όσον αφορά τη μέθοδο εργασία. Είναι απαράδεκτο αυτό και δεν θα ήθελα να επαναληφθεί. Ήρθε το κείμενο, κατόπιν είδαμε ότι κάποιος είχε κάνει λάθος, ήρθε ένα νέο κείμενο και Τελικά μας έμεινε μία μόνο ημέρα για να υποβάλουμε τροπολογίες. Κατόπιν μάθαμε ότι μπορεί κάποιος να υποβάλει τελικά ατομικά τροπολογίες, όχι εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι με αυτές τις συνθήκες εργασίας η συζήτηση δεν μπορεί εύκολα να γίνει. Πέρα λοιπόν από το ότι δεν συμβαδίζει με τους κανόνες, θεωρώ ότι είναι και απαράδεκτο και ελπίζω η Πρόεδρος να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο της πρότασης, ε, έχω και εκεί κάποιες ε, δυσκολίες. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ξεχνάει κατά κάποιο τρόπο στις μελλοντικές της προοπτικές την κοινωνική πτυχή. Βεβαίως δεν είμαστε επί της ουσίας επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας, είναι η οικονομική. Αλλά εν πάση δεν μπορούμε εδώ να παραγνωρίσουμε ότι οι κοινωνικές προτάσεις, οι κοινωνικές πτυχές ε, έχουν παραμεριστεί από το κείμενο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποιες προτάσεις ρεαλιστικές που να έχουν κάποιο περιεχόμενο. Για μένα το κείμενο αυτό δεν ανταποκρίνεται σε αυτήν την προοπτική. Υπάρχουν ε, κάποια μηνύματα, κάποια σλόγγαν, αλλά πολύ φοβάμαι ότι μετά την ψηφοφορία απολύτως τίποτα από αυτά που τελικά θα περάσουν στην ψηφοφορία της Οικονομικής Επιτροπής δεν θα είναι πράγματα που εμείς έχουμε προτείνει. Ποιος τελικά θα συμμετάσχει. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε εμείς να το αποφασίσουμε, μπορούμε απλώς να εκφράσουμε την επιθυμία μας και θα έχει νόημα αν το περιεχόμενο που θα δώσουμε θα είναι ρεαλιστικό. Βεβαίως μπορεί κανείς να μιλήσει για ικανοποιητική αμοιβή ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απλώς μια σύσταση προς τα κράτη-μέλη με σκοπό να φτάσουμε κάποια μέρα σε μια εθνική νομοθεσία που να ανταπεκρίνεται σε αυτές τις επιθυμίες. Αυτό δεν λέγεται όμως κοινωνική πολιτική καθότι αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά έχουν τα κράτη-μέλη. Επίσης υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που δημιουργούν μεγάλα εμπόδια σε μια τέτοια ευρωπαϊκή πρόταση. Εγώ, παραδείγματος χάρη, επισκέφθηκα τη Βουλγαρία και είδα ότι μεταξύ Σουηδίας και Βουλγαρίας υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, τεράστιες διαφορές. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί όταν λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο επίπεδο. Αλλιώς θα πρέπει αυτό το ελάχιστο ευρωπαϊκό επίπεδο να το περιορίσουμε στις χώρες που έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα ε, και προβλεπόμενες αποδοχές. Όσον αφορά τώρα την πρόταση της εισηγήτριας Για το σημείο ένα των συστάσεων θα ήθελα εδώ να πω ότι και εδώ πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και ρεαλιστές. Αλλιώς εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτή την πρόταση. Αυτό που ακούστηκε όσον αφορά τις επιθεωρήσεις εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό είναι αδύνατον. Όχι μόνο επειδή εδώ τα συστήματα στις χώρες είναι διαφορετικά, αλλά και επειδή υπάρχει η αρχή της επικουρικότητας. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερο συντονισμός μεταξύ των εθνικών αρχών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εδώ μια νέα αρχή για την ε, επιθεώρηση εργασίας. Αυτό απλώς θα δημιουργήσει πιο αρνητικές αντιδράσεις ε, προς την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την πράσινη κάρτα, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Ίσως θα πρέπει να την σκεφτούμε λίγο περισσότερο, να την επεξεργαστούμε. Ναι, κάτι τέτοιο θα ήταν μια πολύ καλή πρόταση, την υποστηρίζουμε, γιατί θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε εμείς που εκπροσωπούμε τελικά τους Ευρωπαίους πολίτες, θα έχουμε λίγο περισσότερη δυνατότητα παρέμβασης. Συμβαστική πρόταση G και σύσταση 1, όπως είπα και προηγουμένως, δεν πρόκειται να τις υποστηρίξουμε και θα ήθελα πραγματικά να σας πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από το κείμενο και πιστεύω ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα την καταψηφίσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σέρκας. Πρόεδρε, και εγώ θα κάνω κάποια σχόλια, όπως και συνάδελφος Όρη. Καταρχήν για τη μεθοδολογία και κατόπιν επί της ουσίας, ε, για αυτό που συζητήσαμε και σήμερα το πρωί για τη μεθοδολογία. Έχετε, έχει δίκιο ο κύριος Όρη για να λέει ότι έπρεπε να εργαστούμε στα πλαίσια μιας έκτακτης κατάστασης, αλλά εμένα δεν με εκπλήσει αυτό. Γιατί όσοι εργαστήκαμε για αυτό το φακέλο, ξέρουμε εδώ και τέσσερις μέρες ότι υπήρξε ε, νομοθετική πρόταση πρωτοβουλία και έτσι λοιπόν έπρεπε να τροποποιήσουμε κι εμείς ε, το δικό μας έργο για να είμαστε αποτελεσματικοί. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι καθώς ήταν πάρα πολύ σημαντικό να σεβαστούμε τις προθεσμίες και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε σήμερα τη γνωμοδότησή μας, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι έχουμε τους κανόνες για να μας εξυπηρετούν και όχι το αντίστροφο και έπρεπε κάπως να εργαστούμε σκληρά και το Σαββατοκύριακο, αλλά κάναμε μια χρήσιμη δουλειά και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το έργο των βουλευτών ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν πρέπει να θυσιζόμαστε στον πρόγραμμα των διαδικασιών. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πολύ σημαντικό ο φάκελο αυτό. Ο φάκελο αυτό θα είναι ένα από του πιο σημαντικού στη δική μα ε, θητεία. Είναι το μέλλον τη Ευρώπη και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, γιατί μιλάμε για τροποποίηση των συνθήκων ε, στι εκθέσει του κυρίου Βαν Ποια είναι η αλήθεια, ότι σε όλες τις διαδικασίες που υπάρχουν εδώ, σε όλα τα επίπεδα, ότι αυτή, για αυτή την Επιτροπή ε, είναι η μόνη ευκαιρία να ακουστεί η φωνή της. Έτσι λοιπόν, μιλάμε εδώ για μία εξίσωση που πρέπει να επιλύσουμε. Εμείς ε, θέλουμε να έχουμε φωνή, ε, θέλουμε να ακουστεί η φωνή της Επιτροπής Απασχόλησης στη μεταρρύθμιση που θέτει ο Πρόεδρος Συμβουλίου. Εγώ νομίζω ότι ναι. Και θέλουμε να ακουστεί και δυνατά η φωνή μας και με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Γιατί εμείς τα όσα θα πούμε, κανείς δεν θα τα πει σε αυτό τον Νίκο. Τώρα, για το θέμα που συζητούμε επί της ουσίας, εγώ νομίζω, ε, όσο και αν παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας, βλέπουμε ότι μετά από τρία έτη κρίσης ε, και αφού εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη οικονομική και νομισματική πολιτική, σήμερα στον ισπανικό τύπο, ε, αναφέρεται ότι το 85% των Ισπανών ε, και των ψηφοφόρων ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν συμφωνούν με αυτή την πολιτική η οποία έχει ξεχάσει εντελώ την κοινωνική διάσταση. Ομόφωνα το πιστεύουν αυτό. Όλοι οι πολίτες, κοινωνία λένε φτάνει πια. Γιατί τρία χρόνια μετά σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόστηκε αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι τρία χρόνια πριν και όχι χειρότερα με οποιοδήποτε τρόπο ή λίγο χειρότερα, πολύ χειρότερα είναι μη βιώσιμη η κατάσταση. Υπάρχουν χώρες που πραγματικά κινδυνεύουν να έχουν θεσμικό πρόβλημα, πρόβλημα δημόσιας τάξης. Και ξέρετε θα έχουμε γεγονότα που δεν έχουμε δει τα τελευταία 50 χρόνια στην Ευρώπη. Όμως και τα οικονομικά είναι χειρότερα και είναι χειρότερα γιατί όταν οι πολίτες μας λένε κατά 80% ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε νομίζω ότι εμείς πρέπει να ακούσουμε τι λέει ο λαός εμείς οι βουλευτές και φυσικά με σοφροσύνη, με λογική, αλλά είναι στιγμή μεγάλων αποφάσεων στο κοινοβούλιο αυτό. Και οι μεγάλε αποφάσει στο κοινοβούλιο αυτό είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή πρέπει να έρθει και από εμά και θα πρέπει να βάλουμε στην ημερησία διάταξη του νέου, του ενέργου, γιατί είναι απαραίτητο και δίκαιο. Γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει οικονομική ανάκαμψη αν ε, μειώνουμε την εσωτερική ζήτηση, την κατανάλωση, τι δυνατότητε εκπαίδευση, κατάρτισης, όλα αυτά καταστρέφονται αυτά τα χρόνια στα κράτη-μέλη μας ε, και έτσι δεν θα έχουμε μέλλον, δεν έχουμε παρόν, δεν θα έχουμε μέλλον ούτε οικονομικό μέλλον. Και κλείνω, Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα αυτό που αποτελεί πρόβλημα για ορισμένε ομάδε. Κάποιε αναφορέ μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την πραγματικότητα και να ξεχάσουμε ποια είναι η δική μας ευθύνη. Και η δική μας ευθύνη ότι στο κείμενο του κυρίου Βανέροπον δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για τα κοινωνικά θέματα, για τους νέους στην Ευρώπη, για το τι θα κάνουμε με το δικό μας κοινωνικό μοντέλο. Πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα με τέτοιο τρόπο και να αφήσει ε, να διαφύγει η Επιτροπή αυτή η ευκαιρία. Έτσι λοιπόν σας ζητώ να καταβάλλετε μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να κάνουμε το πιο χρήσιμο. Όμως ε, αυτό το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή δεν μπορεί να σιωπάσουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερο την εμπειρία σας και τη σοφία σας και θεωρώ ότι είστε υπεύθυνο άτομο. Ιδιαίτερα εφόσον ήσασταν πρόεδρος της Επιτροπής Οίκων στην προηγούμενη θητεία. Άρα, όταν προτείνουμε εργαλεία για την έξοδο από την κρίση, πρέπει τα εργαλεία αυτά να είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, να είναι ρεαλιστικά. Νομίζω ότι η μέθοδος εργασίας όμως εδώ ήταν λανθασμένη διαδικαστικά τουλάχιστον, το έχουν πει και άλλοι. Πρόκειται για πολύ σημαντικό έγγραφο που μιλάει για το μέθο, μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις μελλοντικές γενιές. Είναι λοιπόν πολύ ανάρμοστο να συζητάμε αυτό το θέμα τόσο βιαστικά. Καταλαβαίνω ότι πλησιάζουμε σε εκλογές και θα υπάρχει μεγάλη πίεση και ίσως να, μη να διστάζουμε να αναφέρουμε μερικά μη δημοφιλή στοιχεία εδώ μέσα. Αλλά, <clears throat> αλλά λέγω, αυτά είναι κοντόθωρα πράγματα μπορεί να ωφελούν τις εκλογές, την προεκλογική εκστρατεία, αλλά μακροπρόθεσμα θα, είναι, θα μας βλάψουν. Μερικές από τις ιδέες μου βλέπω ότι εδώ αντικατοπτρίζονται με πολύ στρεβλωμένο τρόπο. Εγώ στο κείμενό μου μιλούσα για περισσότερο ενεργούς ανθρώπους στην αγορά εργασίας, αλλά εδώ έχει στρεβλωθεί η ίδια μου η πρόθεση. Και αυτά που προτείνονται τώρα εννοούν ότι δεν θα είναι πιο ενεργοί, αλλά πιο παθητικοί οι πολίτες και θα εξαρτώνται πάλι από κοινωνικές παροχές. Εγώ αποσύρω το όνομά μου από τη δεύτερη μορφή του συμβιβασμού G. Σύρω. Ευχαριστούμε. Χάρκιν. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να επαναλάβω πολλά από αυτά που είπαν κι άλλοι όπως ότι η βιαστική εξέταση μας τα δυσκόλεψε όλα. Δύσκολη εξέβρεση συμφωνιών και συμβιβασμών και όπως είπε και ο κύριος Όρη πρέπει την κοινωνική διάσταση να τη συμπεριλάβουμε οπωσδήποτε. Νομίζω ότι αυτό ζητάνε οι πολίτες. Και συμφωνώ και με τον κύριο Σέρκας. Πριν από μια εβδομάδα στο Δουβλίνο έγινε μια διάσκεψη όπου πήγε ο αρμόδιος επίτροπος και πολλοί τον ρώτησαν τι θα γίνει με την κοινωνική διάσταση και ο κύριος Άντορ διστακτικά είπε ότι δεν προβλέπεται μέχρι τώρα. Η δυσκολία μας λοιπόν εδώ είναι ότι θέλουμε να διατυπώσουμε προτάσεις που να μπορούν να στηριχθούν από την Επιτροπή Εικόν. Το θέμα όμως είναι μέχρι πού θα οθήσουμε τα πράγματα. Μπορεί κανείς να ξεπεράσει όρια, αλλά Αφού είμαστε Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια προσπάθεια. Τώρα χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί χωρίσαμε σωστά τις δικαιοδοσίες μεταξύ χωρών, μελών και ένωσης. Αυτό βοηθάει πολύ το κείμενο, το βελτιώνει και προσωπικά θα έλεγα ότι τα οικονομικά και τα κοινωνικά πρέπει να συνδυάζονται Η πράσινη λεγόμενη κάρτα επίσης είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Σε μερικές χώρες μέλη υπάρχουν συνθήκες που όμως μετά ακυρώνονται, παραβιάζονται κτλ. Οι συνθήκες όπως ξέρετε στη δική μου χώρα πρέπει να εγκρίνονται με δημοψήφισμα και αυτό είναι, δεν είναι πάντα εύκολο. και αυτό διστάζω να προτείνω νέες συνθήκες. Ίσως για αυτή την πρόταση όμως να χρειάζεται. Είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα και τη δέχομαι, αλλά ας μην προσθέσω τίποτα άλλο. Για δε την υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασίας, χαίρομαι επίσης που ζητούμε μια νέα στρατηγική για τις επιθεωρήσεις εργασίας δεν μπορούμε βέβαια να φανταστούμε ακριβώς πώς θα δούλευε κάτι τέτοιο, αλλά φαντα... Συνεχώς γίνεται λόγος για τις μετακινήσεις και βάρδιες των εργαζομένων. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει πολλές προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτό το θέμα φαίνεται ότι είναι λεπτό και άρα μάλλον θα περιμένουμε να ακούσουμε τι θα μας πει η Κομισιόν. Ούτε αυτό είναι άσκημη ιδέα. Τέλος, όταν μιλάμε για αξιοπρεπείς μισθούς και έσοδα και αποφυγή της ανέχειας και τέτοια, χρειάζονται εδώ με ορισμένοι σταθεροποιητικοί παράγοντες της οικονομίες. Γίνεται λόγος για σύγκληση, αλλά αυτό δεν αρκεί. Το θέμα δεν είναι μόνο η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και άλλους οικονομικούς σταθεροποιητικούς παράγοντες. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπενιόν και μετά ο κύριος Θωμάς Μάν. Μάλιστα. Το θέμα των εργασιακών επιθεωρήσεων με ανησύχησε κάπως γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο τέτοιο πράγμα Έχουμε επιθεωρητές για υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασίας, αλλά όχι επιθεώρηση καθεαυτήν, design επιθεώρηση. Επίσης και σε άλλες χώρες μέλη νομίζω ότι άλλες έχουν τις α δομές και άλλες τις β. Άλλα ονόματα έχουν σε μία χώρα, άλλα στην άλλη κλπ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί του συμβιβασμού συμπεριλάβατε τις περισσότερες μου ντροπολογίες. Έχω όμως ακόμη ένα πρόβλημα. Ξέρω ότι η συνάδελφος Μάριον εδώ πέρα μίλησε για το θέμα του ελαχίστου εισοδήματος, αλλά δεν γνωρίζω στα πλαίσια του κειμένου αυτού τι θα μπορούσε να εννοεί κάτι τέτοιο, τι είναι εισόδημα. Μπορεί να εννοεί πολλά πράγματα. Ο κύριος Ορή φοβάται ότι μπορεί να είναι ενιαίο πανενοσιακό ελάχιστο εισόδημα, πράγμα το οποίο δεν θα ήταν και πολύ πρακτικό, ελπίζω να μην εννοεί αυτό. Μίσος εννοεί αντίθετα απλώς την ενθάρρυνση των χωρών μελών να καθορίσουν δικές τους μεθοδολογίες για το δικό τους ελάχιστο εισόδημα. Αυτό θα ήταν αποδεκτό. Μεταξύ των δύο ακραίων αυτών θέσεων θα μπορούσε να υπάρχει και μία λίγο πολύ ε, κάποιος τύπος που να λέει ότι μπορεί να μην καθο... χρειάζεται να καθορίσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κάθε κράτος τον ελάχιστο μισθό αλλά όποιο και να είναι το ελάχιστο εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνάει το ΑΕΠ, το σύνολο. Ως προς τα άτομα τι σημαίνει ε, ελάχιστο εισόδημα, εννοεί ζεύγη, νοικοκυριά, θα αλλάζει ανάλογα με το αν έχουν παιδιά ή όχι, θα είναι ατομικό. Θα αλλάζει για τις πολύτεκνες οικογένειες θα ξεπερνάει αυτά που μπορεί να αναμένει κάποιος να κερδίζει από μια κανονική μικροαστική θέση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν ξέρω τι εννοεί κατώτατο εισόδημα. Ούτε καν εισόδημα τι εννοεί. Ευχαριστώ. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Θωμάς Μάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ανήκω και στις δύο αυτές επιτροπές. Είμαι αντιπρόεδρος εδώ, αλλά ανήκω και στην οικονομική. Γνωρίζω λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια τη θέση των μεν και των δε. Έχετε δίκιο. Πρέπει να δούμε πώς στο τέλος θα είναι ισορροπημένη η πρόταση που θα κάνουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να γίνει αυτό. Στην Ισπανία σήμερα ο κόσμος είναι στους δρόμους, διαδηλώνει. Και το ερώτημα είναι, εμείς από τη Γερμανία θέλουμε να καταλάβουμε πώς ε, οι προτάσεις που θα κάνουμε για τη μείωση των λιμάτων θα είναι λογικές. Απ' την άλλη χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια δημοσιονομική ένωση. Για να γίνει αυτό χρειάζονται πρωτοβουλίες και μείωση των διαφορών και του χάσματος. Και εγώ μίλησα και με Έλληνες. Αύριο ξέρετε ότι πάει στην Αθήνα η Άγγελα Μέρκελ. Και προσπαθήσαμε να μην γίνει η αυριανή ημέρα μία μέρα όπου απλώς θα υπάρχουν διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Χρειαζόμαστε κάτι που να μην μοιάζει με απέτηση και επιβολή από τα πάνω προς τα κάτω. Να υπάρχει μια ισορροπημένη προσέγγιση, μια σωστή προσέγγιση, να υπάρχει προοπτική για αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Αν αυτό το περάσουμε σαν εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, θα έχουμε κερδίσει. Και βεβαίως πάντα προσπαθούμε να φτάσουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις με ευελιξία και ξέρω ότι πολλές φορές οι χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλιστές μπορούν να συμφωνήσουν. Εδώ βλέπετε η πρόθεση της κυρίας Μέρκελ είναι καλή. Ελπίζω το μήνυμα που θα περάσει να είναι θετικό. Το θέμα τώρα του ελάχιστου εισοδήματος, των ελάχιστων ε, αποδοχών. Εδώ φυσικά και θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει στην κάθε περιφέρεια, στην κάθε χώρα, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων βεβαίως και ανάλογα με την παράδοση και την ομοθεσία της κάθε χώρας. Και βεβαίως το βασικό είναι ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν να επιβιώσουν. Οι διαφορές υπάρχουν, αλλά το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε προς τα έξω είναι ότι δεν θέλουμε περισσότερους αποκλεισμούς, περισσότερες διαφορές. Δεν θέλουμε να υπάρξουν χαμένες γενιές. Όχι. Όχι. Αυτό χρειαζόμαστε, μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά εδώ την νομισματική και οικονομική ένωση. Κοιτάξτε, εδώ είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι μπορούμε να προοδεύσουμε. Το έγγραφο, κυρία Πρόεδρε, είναι καλό. Βεβαίως υπάρχουν σημεία τα οποία θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω. Η κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο. Ξέρω ότι έχουν συμμετάσχει οι συνάδελφοι από την ομάδα μας στην συμβαστική πρόταση. Όσον αφορά το ελάχιστο όμως εισόδημα, εδώ έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ εκφράζει αντιρρήσεις, αλλά υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα ελάχιστο εισόδημα. Και το πιο σημαντικό για μας εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο είναι ότι ο τρόπος που καθορίζονται αυτά τα ελάχιστα εισοδήματα, οι ελάχιστες αποδοχές, θα πρέπει να οδηγήσουν τα κράτη-μέλη να μην ξεπερνούν ένα κατώτατο όριο. Και βεβαίως, όταν μιλάμε για αξιοπρεπές ε, εισόδημα, ελάχιστο εισόδημα, εννοούμε κάτι που επιτρέπει σε έναν Ευρωπαίο πολίτη να ζήσει με αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι το ζητούμενο τελικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, για τους περισσότερους από εμά. Γι' αυτό και κάποια από τα κριτήρια που προτείνονται εδώ θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το πακέτο για την νομισματική ένωση. Είτε μας αρέσει η έννοια της νομισματικής ένωσης ή όχι. Η κοινωνική διάσταση είναι εξαιρετικά σημαντική. Και Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε και λίγη κοινωνική πτυχή. Όπως ξέρετε είναι τελείως διαφορετικό το επίπεδο της κοινωνικής προστασίας από τη μια χώρα στην άλλη. Υπάρχουν και περιπτώσεις των διασυνοριακών συμφωνιών. Το θέμα τώρα των δικτών που έχουν συμπεριληφθεί εδώ που χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η ποιότητα ζωής. Αυτό βέβαια πρέπει να ξεπερνάει το ΑΕΠ. Και εδώ έχουμε συνεργαστεί και με το ε, Διεθνές Γραφείο Εργασίας για να θεσπιστούν αυτοί οι ε, δείκτες. Ο Τόμας Χάντελ έχει το λόγο. Κοιτάξτε, ακούγοντας ε, τους μεν και τους δε, συνειδητοποίησα ότι ένας γνωστός συγγραφέας Ευρωπαίος είχε γράψει ότι θα ήταν ίσως καλύτερα με τη σιωπή να ξεπεραστούν κάποιες αμφιβολίες παρά κάθε φορά να προσπαθεί να πείσει με την αντιπαράθεση και τα επιχειρήματα. Για το θέμα του ελάχιστου εισοδήματος. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στο σχέδιο έκθεσης της εισηγήτριας αναφέρεται ότι αυτό θα πρέπει να είναι το 60% του μέσου εισοδήματος μιας χώρας. Αυτό ήταν στην έκθεση της εισηγήτριας σαν πρόταση. Για την κάθε χώρα λοιπόν βλέπουμε ότι το ελάχιστο εισόδημα θα πρέπει να οριστεί σε σχέση με τα δεδομένα της κάθε χώρας. Με αυτό εννοείται δεν μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε για ευρωπαϊκό ε, μέσο όρο και πρέπει να βασιστούμε στα κριτήρια του ΟΣΑ για το πότε ξεκινάει αυτό το επίπεδο κάτω από το οποίο ξεκινάνε οι συνθήκες ε, μη αξιοπρεπούς ε, διαβίωσης και παινίας. Αυτό το 60% λοιπόν του μέσου εισοδήματος μιας χώρας είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να βασιστούμε. Σήμερα βλέπουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ανησυχίες και φόβοι για το μέλλον. Ο κόσμος εγκαταλείπει την Ευρώπη λόγω αυτών των φόβων και των ανησυχιών. Και όταν μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης και τις προπτικές και ακούμε τον Πρόεδρο Μπαρόζο, βλέπουμε ότι αυτό που σίγουρα θα πρέπει να μας απασχολήσει εμάς είναι ποια κριτήρια θα ορίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε αυτή η κοινωνική Ευρώπη να μην αποδυναμωθεί ακόμα παραπάνω. Και αυτό το ελάχιστο εισόδημα, αυτές οι ελάχιστες αποδοχές, σίγουρα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα κριτήρια. Σήμερα αναφερόμαστε σε 27 κράτη-μέλη της Ευρώπης, όπου δύο δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του ελάχιστου εισοδήματος. Κάτι λοιπόν θα πρέπει εδώ να υποβάλουμε σαν πρόταση στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Αλλά και κάτι άλλο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Κάτι δεν μπορώ να το δεχτώ. Μονίμως επικαλούμαστε την ε, επικουρικότητα όταν κάτι δεν μας αρέσει. και εδώ άκουσα τον συνάδελφο Όρη. Όταν μιλάμε για τις ελάχιστες αποδοχές, όταν αναφερόμαστε στις συνθήκες εργασίας ναι. και πολλά άλλα, και πολλά άλλα στοιχεία. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αν θέλουμε να ενδυναμώσουμε την κοινωνική Ευρώπη. Γιατί αν η εντύπωση που δίνουμε είναι ότι αυτοί που αποφασίζουν στην Ευρώπη δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις ανησυχίες, τότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι και ότι οι ανησυχίες των Ευρωπαίων διαρκώς θα αυξάνονται. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι εδώ έχουμε μια έντονη συζήτηση γιατί πρόκειται για ένα θέμα αρκετά λεπτό. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και όλοι γνωρίζουμε ότι η κοινωνική διάσταση είναι πολύ σημαντική. Και επίσης ε, μπορεί και από ιστορική σκοπιά να είναι καθοριστική σημασία. Όμως, εγώ έχω την ακόλουθη άποψη λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση Tyson, ίσως θα είχε περισσότερο νόημα το ζήτημα αυτό να είναι αντικείμενο ξεχωριστής έκθεσης, αντί να το συνδέουμε με άλλο θέμα. Και ξέρουμε ότι η αρμόδια επιτροπή δεν θα μας οδηγούσε στα επιθυμητά αποτελέσματα σε... για κάποια από τα στοιχεία που ακούστηκαν στη συζήτηση δεν συμφωνούμε. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε μία σειρά αρμοδιοτήτων και κάποιες αρμοδιότητε δεν τι έχουμε. Αυτό βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. η οποία καθορίζει μία σειρά αρμοδιοτήτων, όμως έχουμε και εμεί αρμοδιοτήτων που μένουν εκτό Θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε εδώ να θέσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό, ένα νούμερο, αλλά γνωρίζουμε ότι ακόμη και αν εδώ λέγαμε ότι το 45% του ενεργού πληθυσμού πρέπει να εργάζεται, Όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, ακόμη και αν εμφανίζεται σε κάποια νομοθεσία. Και να εκπονούμε νομοθεσία που δεν μπορεί να τη θέσει εφαρμογή είναι κάτι εντελώ άχρηστο. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να μιλήσουμε για το ελάχιστο εισόδημα, σε αυτό συμφωνώ. Όμως ε, υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά επιδόματα. και τα δίκτυα κοινωνική στήριξης. Έτσι λοιπόν, ε, να μιλάμε για μια νέα ευρωπαϊκή εστίαση ή για μια ομοιόμορφη στήριξη στους ευρωπαίους ενέργους. Ουσιαστικά θα ήταν υπερβολική εμπλοκή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν, παραδείγματο χάρη, πάρα πολλέ διαφορέ σε ό,τι αφορά τι άδειε μητρότητα. Τα κοινωνικά συστήματα διαφέρουν πάρα πολύ και να το θέτουμε εδώ και να θέσουμε κάποιου κοινού όρου μπορεί να φαινόταν απλό καταρχήν, αλλά στην ουσία δεν είναι. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Υπάρχουν πάρα πολλέ συμβαστικέ τροπολογίε εδώ και πολλέ θα εγκριθούν αύριο. Αυτό είναι βέβαιο όμω. Ορισμένα ζητήματα είναι προφανές ότι έχουμε αποκλήσει ε, απόψεων. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά το εξής. Στην τελευταία ε, θητεία προσπαθήσαμε να έχουμε ένα νομοθετικό κείμενο με την κυρία Λάμπερτ όπου θα συμπεριλαμβανόταν η ιδέα πως ε, θα έπρεπε να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός συντονισμός των επιθεωρήσεων εργασίας. Δηλαδή να μην ε, έχουμε έναν φορέα ευρωπαϊκό, όπως λέει σήμερα η πρόταση, αλλά να έχουμε συντονισμό. Και δεν το καταφέραμε. Διαφέρει η σημερινή κατάσταση, αυτό είναι αλήθεια. Όμως δεν υπάρχει νομική βάση για να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. θα πρέπει να αεροβατούμε. Θα πρέπει να προτείνουμε μέτρα που μπορούν στη συνέχεια να γίνουν πραγματικότητα. Και να αποφύγουμε στη συνέχεια να ξεχαστούν οι δικές μας ιδέες στην Αρμόδια Επιτροπή γιατί δεν θα ανταποκρίνονται στο κύριο θέμα που μας απασχολεί. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούγοντας τη συζήτηση, παρατηρεί κανείς δύο πράγματα. Από τη μία τα οικονομικά και οι δοσοληψίες, απ' την άλλη η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ακούν και οι συνάδελφοι όταν πηγαίνουν στην εκλογική τους περιφέρεια. Κατανοώ ότι μπορεί οι λαοί όπως στην Ισπανία να μην δέχονται πια τα μέτρα λιτότητας που τους επιβάλλονται. Απ' την άλλη όμως στη Γερμανία επίσης ο κόσμος μου λέει μα και σε εμά γίνονται εξοικονομήσεις και σφίγγουμε το ζωνάρι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει γενικότερα έλεγχος. Καταλαβαίνετε τους δε και το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να επιδειχτούμε μανιχαϊστέ και μανιχαίστριες. Πρέπει να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Όχι μόνο στην Επιτροπή μας αλλά και σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Να ακολουθήσουμε την μέση οδό. Το λυπηρό είναι ότι ο όρος κοινωνική διάσταση έχει γίνει πια σύνθημα κενό. Οι μεν το απορρίπτουν τελείως, οι δε το υποστηρίζουν μέχρι θανάτου. Πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο τον όρο αυτόν. Να δούμε τι κοινωνικά μέτρα πρέπει και μπορούν να ληφθούν, λογικά, κάποια εγγύηση για τους νέους δηλαδή και Επίσης κοινωνικά μέτρα, υπάρχουν κοινωνικά μέτρα που ίσως δεν δικαιολογούνται πια, είναι εκλογικά ή προεκλογικά ή μετεκλογικά δώρα και πρέπει να προσέξουμε να μην τα βλέπουμε όλα άσπρο μαύρο. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την βιωσιμότητα και να προσιλωθούμε στο μέλλον. Τώρα, ελάχιστο εισόδημα ή μισθός. Νομίζω ότι το ελόχιστο εισόδημα δεν είναι μόνο ένας μισθός. Είναι γενικά ότι χρήματα διαθέτει κανείς. Στα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχει ένα σύστημα περίθαλψης που εγγυάται κάποιον μισθό. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει, πρέπει να συζητηθεί ακόμη το θέμα του κατώτατου μισθού. Μπορεί να υπάρχουν επίσης αδικαιολόγητοι μισθοί, αλλά ένα κατώτατο εισόδημα που να εγγυάται την επιβίωση των πάντων, αυτό είναι κάτι σωστό. Σιπέλ μήπως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν σκοπεύω να ζητήσω το λόγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, όμως άκουσα κάποια πράγματα και να ρωτιέμαι αν κάποιοι συνειδητοποίησαν ε, που ζούμε και ότι εδώ βρισκόμαστε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το θέμα του του μισθού δεν ε, συζητείται μόνο εδώ και δύο χρόνια, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. ουσιαστικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από το μηδέν για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά τώρα δεν υπάρχει χρόνος, δεν έχει νόημα να ξεκινήσουμε ε, και πάλι τη συζήτηση από το μηδέν, γιατί ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και δεν έχουμε χρόνο. Ο κόσμος θέλει λύσεις στα προβλήματα που έχει η Ευρώπη τώρα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πολύ διαφορετικά προβλήματα από αυτά που αναφέρονται δημοσίως. Κάποιοι αναρωτιούνται αν ε, η Γερμανία θα πρέπει να κάνει τα πάντα ή αν θα πρέπει να πληρώσει τα ελληνικά χρέη. Και ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ε, και προβλήματα με τα κόμματα και εμεί προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις. Ε, Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν άνθρωποι που του έχουν μειώσει τι συντάξει και δεν μπορούν να ζήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που στο τέλο τη ημέρα θα πρέπει να ζητήσουν ε, από ε, την ε, κυβέρνηση επίδομα γιατί τελικά δεν τους φτάνει ο μισθός να ζήσουν. Έτσι λοιπόν, ακριβώς εδώ, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, θα πρέπει εμείς να επιζητήσουμε λύσεις γρήγορα και όχι να μπαίνουμε σε τέρμονες συζητήσεις. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να επιβιώσει κάποιος ε, με όσα κερδίζει από την εργασία του. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, πολύ σύντομα, θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με τη διαδικασία αυτή. Ο τρόπος ε, που καταρτήσαμε αυτή την γνωμοδότηση δεν με ικανοποίησε καθόλου ούτε σεβαστήκαμε καθόλου τους κανόνες που έχουμε. Και αναρωτιόμουν αν ε, πρόκειτο να συνεχίσουμε τη διαδικασία αυτή και με άλλες εκθέσεις. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Μπάουερ. Αν ήμασταν ε, κάπως πιο μετριοπαθείς με την εκθέση αυτή, ίσως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και τις δικές μας απόψεις στο τελικό κείμενο. Γιατί τώρα έχουμε υιοθετήσει κάποιες ακραίες απόψεις για τις οποίες δεν μπορούμε να βρούμε υποστήριξη. Και εγώ θεωρώ ότι οδηγούμαστε σε αποτυχία. Ευχαριστώ για αυτή την ε, πλούσια συζήτηση, λέει η Πρόεδρος. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια καταρχήν και πάλι επί της διαδικασίας και επί του τρόπου που μπορούμε να συμμετέχουμε εμείς στη συζήτηση αυτή. Όλοι γνωρίζουν ότι ο κύριος Φαρουπό υπήρε την ε, πρωτοβουλία για τη συζήτηση αυτή και είναι μια συζήτηση που γίνεται κυρίως στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στη συζήτηση έτσι όπως θα υλοποιηθεί το Δεκέμβριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορες δομές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι απολύτω νόμιμο και γιατί είναι σημαντικό να τοποθετηθεί και το Κοινοβούλιο με τη δική του φωνή πριν αυτή η τόσο σημαντική συζήτηση να λάβει χώρα το Δεκέμβριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα υλοποιηθεί με ένα ρυθμό ανεξαρτήτως του δικού μας. Ακούσαμε τον πρόεδρο Μπαρόσο, ακούσαμε ότι στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ανέφερε τη δική του θέση, παρουσίασε τη δική σου θέση και παρουσίασε ποιο είναι ο χαρτής πορείας κατά την άποψή του. Κατόπιν ε, είδαμε το έγγραφο που παρουσίασε ο πρόεδρος Φαν σε τέσσερα μέρη, δεν συμπεριλαμβάνεται και η κοινωνική πτυχή για να ξεκινήσει η συζήτηση το Δεκέμβριο. Και εγώ νομίζω ότι όλοι εδώ γνωρίζουν το έργο που υλοποιεί ο κύριος Βεστερβέλε μαζί με κάποια κράτη-μέλη. Παράλληλα. Κοιτάξτε εδώ, δεν θα συζητήσουμε τι θέλουμε στον ιδανικό κόσμο, αλλά εδώ πρέπει να δούμε πώς το συγκεκριμένο πλαίσιο οι ανησυχίες ε, που μας απασχολούν εδώ, σε αυτή την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και εγώ πολλές φορές ε, αισθάνθηκα μεγάλη συνένεση σε αυτό το θέμα από την δική μας Επιτροπή. Πώς λοιπόν αυτές τις ανησυχίες ε, θα τις συμπεριλάβουμε σε συζητώνται σήμερα. Σε ένα πλαίσιο, και το υπενθυμίζω, είναι το εξή. Ζούμε σε μία κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είναι η σπονδυλική στήλη του συστήματος των οικονομικών πολιτικών δηλαδή μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Σε ένα νομικό πλαίσιο, όπου μια, όπου μια μεγάλη πρόοδος ε, που υλοποιήσαμε ήταν η οθέτηση μιας χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνει και μια πολύ σημαντική κοινωνική επιτυχία και μια αναθεώρηση της συνθήκης της Λισαβόνας περιλαμβάνει το άρθρο 9 και ουσιαστικά καθιστά το κοινωνικό ζήτημα οριζόντιο και το περιλαμβάνουμε κάθε φορά. Παρεμβαίνουμε σε ένα πλαίσιο όπου αυτό που διακυβεύεται ουσιαστικά είναι η δεύτερη περίοδος της ΟΝΕ όταν μιλάμε για την ΟΝΕ, έχουμε πάντοτε την ε, πεποίθηση, την εντύπωση ότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ τη οικονομία και του νομίσματο. Όμω, αν δείτε τι συνέβη, όταν μπήκαμε στο ευρώ, όταν εθετήσαμε τη συνθήκη του Μάστρικτ, όταν εθετήσαμε τα εργαλεία τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση, υπήρχε μια ισορροπία στην οποία Αναφερόμαστε πάντα στο άρθρο 129 για τις οικονομικές πολιτικές και το άρθρο 148 για τις κοινωνικές πολιτικές. Αυτή η ισορροπία όμως δεν είναι ικανοποιητική. Αλλά αν ε, εμείς, ε, η δική μας Επιτροπή, δεν πει τίποτα, τότε αυτή η ισορροπία που δεν είναι και ιδιαίτερα ικανοποιητική θα καταστραφεί υπό την πίεση των κύριων πρωταγωνιστών, δηλαδή των οικονομικών ε, φορέων, των φορέων των χρηματογορών. Εγώ Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κυρία Μπάουερ. Και κάποιοι θα το θυμούνται. Όταν ε, ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, βάσει αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προτάσεις του κ. Φαρουμπάη, εγώ ήθελα να εκπονήσουμε εμεί τη δική μας έκθεση και το ζητήσαμε αυτό να εκπονήσουμε τη δική μας έκθεση. Όμω ε, υπήρχε αντίρρηση από την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Και εμείς ζητήσαμε ενισχυμένη συνεργασία. Και μόνο η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ε, επί του παρόντος ε, μπόρεσε να πετύχει αυτή την ενισχυμένη συνεργασία. Επομένως, δεν ε, είχαμε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση για να μπορέσουμε να καθορίσουμε το δικό μας χρονοδιάγραμμα και να καθορίσουμε τα δικά μας εργαλεία. Πρέπει να προσαρμοστούμε, όσα υπήρχαν επιτάπητος Κοιτάξτε, δεν λέω ότι πρέπει να τρέχουμε πίσω από τους άλλους, γιατί το μισό αυτό, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά που είναι διατέθημα για να μπορούμε να λέμε κάποια πράγματα. Και αύριο το απόγευμα έχω ραντεβού με την κυρία Τάισεν, έτσι ώστε αμέσως μετά την ψηφορία στη δική μας επιτροπή να μπορέσουμε να συζητήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς τις ανησυχίες που εξέφρασε ο κύριος Όρη. Δηλαδή να υποστηρίξουμε προτάσει που και η κυρία Τάισαν θα μπορούσε να εντάξει στη δική τη έκθεση και είχα ήδη τη δυνατότητα να συζητήσω μαζί της. Και ο κύριος ε, Τόμας Μάν συμμετέχει και στις δύο επιτροπές. Έτσι λοιπόν, εμείς ε, θέλουμε να επαναφέρουμε την ισορροπία στην πρόταση, αλλά συζήτηση είναι ανοιχτή. Δεν ξέρω ακόμη ως πού θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή τη συμφωνία. Τώρα, για τις διάφορες ανησυχίες που εκφράστηκαν από εσά. Για το αν τα κοινωνικά δικαιώματα που διεκδικούμε ε, είναι κοινωνικά δικαιώματα σε επίπεδο όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν θα επιβάλλουμε ελάχιστο μισθό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κυρία Χάρκιν, ορθά υπογράμμισε ότι στο συμβιβασμό, στο συμβιβασμό G και στη σύσταση 1 κάνουμε τη διάκριση μεταξύ μιας πολιτικής της Ένωσης, αυτού που πρέπει να είναι πολιτική της Ένωσης και αυτού που προκύπτει από το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας, δηλαδή της παρακολούθησης, της παράλληλης παρακολούθησης των δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των όσων άπτονται της αρμοδιότητας των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου και του μισθού. Εγώ ποτέ δεν άκουσα κανένα να προτείνει έναν ενιαίο κατά του μισθό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Και αν μιλάμε για κάτι τέτοιο, δεν θέλουμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Αλλά διαπιστώνω ότι το Συμβουλίο της Ευρώπης το ίδιο έχει κάνει, ε, έχει θέσει το 60% ε, του μισθού ως κατώτατο μισθό σημείο αναφοράς. Και το αναφέρει ο κ. Χέντελ αυτό. Έχουμε μια αρκετά πολύπλοκη διατύπωση, αλλά δεν παραπέμπει ακριβώς ρητά σε έναν κατώτατο μισθό, γιατί τι προτείνεται. Στο πλαίσιο ε, και των ερμοδιοτήτων κρατουμένων αξιοπρεπείς μισθούς με ελάχιστα εισοδήματα που να αποτρέπουν την ανέχεια. Έτσι λοιπόν, ε, νομίζω ότι σε αυτήν την έντονη συζήτηση που είχαμε, δεν καλύπτεται ακριβώ η πραγματικότητα των όσων προτείνεται ως συμβιβαστικές λύσεις αύριο. Και εγώ ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Κυρία Χάρκιν, εξέφρασε κάποιες ανησυχίες. Δεν είναι εδώ βέβαια, ελπίζω να τις θα μεταβιβάσουν οι συνεργάτες της ε, για το θέμα της ε, πράσινης κάρτας. Δεν ε, θα υπάρχει αναθεώρηση των συνθηκών. Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι από μια χώρα που ακριβώ ίδια ήταν η κατάσταση και μάλιστα ο πρόεδρο Μπαρόζο και στην ομιλία του για την κατάσταση τη Ένωση είπε ότι η δυνατότητα άμεση αναθεώρηση της συνθήκης ε, δεν πληρούνταν μάλλον. Έτσι λοιπόν, ε, θεωρώ ότι υπάρχει εδώ συνένεση από όλε τι ομάδε και χαίρομαι γι' αυτό. Μία από τις παραγράφου που σας πρότεινα υπενθυμίζει ότι δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως τη δυναμική που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνα σε διάφορους τομείς. Όμως ε, η συζήτηση που θα λάβει η χώρα το Δεκέμβριο είναι μια συζήτηση όπου όλα θα τεθούν επιτάπητο και αν υπάρχουν προτάσεις που εμεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναφερθούν και να συζητηθούν, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τις συζητήσουμε τις προτάσεις αυτές. Και κάτι ακόμη για την κυρία Σάια, για την ε, μεθοδολογία επί της διαδικασίας. Οι περισσότερες τροπολογίες που κατατέθηκαν, κατατέθηκαν από τους κέντες εισηγητές. Εκτός από αυτή την τροπολογία που κατατέθηκε από την κυρία Βλέσης και Και δύο που κατατέθηκαν από εσά. Και όταν συναντηθήκαμε με το σύνολο των σκιωδών εισηγητών, λάβαμε υπόψη την κατάσταση αυτή για να ζητήσουμε υπεύθυνοι των ομάδων να μπορούν να λάβουν υπόψη τι τροπολογίε που είχαν κατατεθεί μεμονωμένα, από συναδέλφους μεμονωμένα. Ο κύριος ε, Σέρκας ε, επανέλαβε κάποιε τροπολογίες του κύριου Πριώτο και ε, Επίση, ε, συμπεριλήφθησαν και κάποιε προηγούμενε προτάσει του κυρίου Όρη. Σε ό,τι αφορά τώρα τι δικέ σα τροπολογίε, είχαν ε, ιδιαίτερη μοίρα γιατί όσες δεν καλύπτονταν από άλλες τροπολογίες θα επανεισαχθούν στον κατάλογο αύριο και κάποιες ρητός έχουν αναφερθεί στους και έχουν συμπεριληφθεί στους συμβασμούς. Ξέρω ότι δεν είναι ιδανική διαδικασία, το αναγνωρίζω, ελπίζω ότι συλλογικά θα δεσμευτούμε να μην το θεωρήσουμε αυτός προηγούμενο, αλλά ως εξαίρεση και ζητώ συγγνώμη γιατί φέρω μεγάλη ευθύνη Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ψηφοφορία αύριο που θα επιτρέψει στην δική μας Επιτροπή να υιοθετήσει μια γνωμοδότηση που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και να επηρεάσουμε τη συζήτηση στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Απέναντι στην κυρία Τάισεν που ξέρω ότι είναι πολύ θετική. Ακούει τις δικές μας ανησυχίες. Σας ευχαριστώ για την ποιότητα της συζήτησης που είχαμε. και στο στάδιο αυτό τη παρουσίαση συμβαστικών τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε αύριο το κείμενο αυτό για να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα τη Επιτροπή ΕΚΟΝ. Τώρα, φτάνουμε στο σημείο έκθεση, έκθεση της κυρίας Μπλίντσεκ Βιτσιούτε σε σχέση με το πρόγραμμα Εράσμους για όλους. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σκιώδη εισηγητή, τους σκιώδης εισηγητές, γιατί μπορέσαμε να συνεργαστούμε πολύ καλά ανταλλάξαμε απόψεις και βρήκαμε και συμβαστικές προτάσεις για πολλά από τα θέματα. Μπορέσαμε να προετοιμάσουμε 34 συμβαστικές ε, τροπολογίες και θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για σκιώδεις εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων συμβιβαστικές τροπολογίες που τελικά υποστηρίχθηκαν από όλους. Θα σας αναφέρω την τροπολογία του Μάρτιν Κάσλερ. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται. Θα ήθελα εδώ πραγματικά να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα που βασίζεται στην διαβίου κατάρτιση και στους ηλικιωμένους. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα, υποπρόγραμμα θα έλεγα, που αναφέρεται σε αυτά τα άτομα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τους ηλικιωμένου και τη δραστηριότητά τους στην κοινωνία, ιδιαίτερα σήμερα, ενώ βλέπουμε ότι η γύρανση του πληθυσμού είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες μας. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην εκμάθηση, στην κατάρτιση των ενηλίκων. Το συζητήσαμε αυτό με τους σκιώδεις εισηγητές και θελήσαμε να καθορίσουμε μία ηλικία όσον αφορά αυτήν την κατάρτιση που αφορά τους ε, ενήλικες έτσι ώστε να καθοριστεί ένα όριο ηλικίας το οποίο να είναι αποδεκτό για όλα τα κράτη-μέλη. Σήμερα το κάθε κράτος έχει διαφορετική ε, θέση όσον αφορά τον καθορισμό της ε, ηλικίας. Άλλοι θεωρούν ότι είναι 18 ετών, άλλοι 20 και κυρίως άτομα τα οποία θα πρέπει να είναι μέχρι 64 ετών. Θεωρώ ότι αυτό το ανώτατο όριο θα πρέπει να εξαλειφθεί, έτσι ώστε να μπορούν άτομα πιο ηλικιωμένα να υποφεληθούν και να υπάρξει πραγματική ε, κατάρτιση και σε άτομα που έχουν ξεπεράσει, παραδείγματος χάρη του 64ου έτους ηλικίας το ελάχιστο όριο ηλικία ε, βεβαίως πρέπει κάπως να καθοριστεί και αυτό το συζητήσαμε με τους ε, σκιώδες εισηγητές και είπαμε ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ανώτατο όριο. Τα κράτη-μέλη έχουν την παράδοσή τους, θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ευέλικτοι και να σεβαστούμε την ε, εθνική παράδοση και εμπειρία. Τώρα, όσον αφορά τις άλλες συμβαστικές τροπολογίες, συμφωνούμε και ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που υποστήριξαν αυτές τις προτάσεις. Όσον αφορά τους νέους, Οι προτάσεις ε, στηρίχθηκαν από όλους τους συναδέλφους. Για τις άλλες τροπολογίες Θελήσαμε να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στο πρόγραμμα, ιδιαίτερα για άτομα με ειδικέ ανάγκες, άτομα με δυσκολίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και η Επιτροπή μας θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Οι σκιώδεις εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων συζήτησαν επίσης ε, για θέματα χρηματοδότησης, προϋπολογισμού αυτού του προγράμματος και συμπεριλάβαμε στις συμβαστικές ε, τροπολογίες την πρόταση για τους διάφορους τομείς η χρηματοδότηση αυτών των ε, προγραμμάτων σίγουρα δεν θα πρέπει να μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Για κάποια προγράμματα προτείναμε μάλιστα αύξηση της χρηματοδότησης και οι σκιώδεις εισηγητές γνωρίζουν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ δυναμικοί όσον αφορά τις προτάσεις μας στον προϋπολογισμό και δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτό τον τομέα στα χέρια μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους τους σκιώδεις συγητές με τους οποίους συνεργάστηκα με πάρα πολύ καλό τρόπο και ελπίζω αύριο στην ψηφοφορία θα υπάρξει ευρεία υποστήριξη αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπακ που είναι, που είναι, να τους, να τους, Δεν κάθεται στη συνήθη θέση του, γι' αυτό δεν τον είπα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Μάρτιν, μάλλον να ζητήσω συγγνώμη διότι ο Μάρτιν Κάσλερ δεν μπορεί να είναι παρόν μου. Ζήτησε λοιπόν να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Ευχαριστεί ιδιαίτερα την εισηγήτρια για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν στην επεξεργασία αυτού του κειμένου. Είναι πολύ σημαντικές οι τροπολογίες που καταφέραμε να υποβάλουμε, οι συμβιβαστικές τροπολογίες το θέμα της διαβίου κατάρτισης είναι εξαιρετικά σημαντικό στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ όλες τις πολιτικές ομάδες που δέχτηκαν τις προτάσεις μου όσον αφορά και τους, πιο ηλικιωμένους. Και θα ήταν τελείως παράλογο να μιλούμε για διαβίου κατάρτιση χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις φάσεις της επαγγελματικής ζωής. Θέλω πραγματικά να πω ότι το θέμα των ε, ηλικιωμένων είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και δίνουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι πραγματικά θα πρέπει εδώ να ενδυναμώσουμε όλες τις προτάσεις για την κατάρτιση, για τη διαβίου κατάρτιση, κατάρτιση των ανηλίκων μέσω του προγράμματος Εράσμους για όλους. Επίσης θα ήθελα εδώ πραγματικά να υποστηρίξω μία από τις προτάσεις μου που δεν καλύπτονται από τις συμβαστικές τροπολογίες. Το θέμα του ονόματος. Έρασμους για όλους. Η πρόθεση εδώ δεν είναι βεβαίως ε, κάτι που φαίνεται από το όνομα αυτό, από τον τίτλο αυτό «Έρασμος για όλους». Και γνωρίζω ότι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπής έχει ήδη δύο προτάσεις για όνομα. Γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να προτείνω την υποστήριξη των τροπολογιών 86 και 87. Θα ήθελα να μιλήσω για τον τίτλο που αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στην γενιά της Ευρώπης, που δίνει έμφαση στην ε, κατάρτιση για όλους. Θα πρέπει να βρούμε ένα τίτλο, ένα όνομα που να μπορεί να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες με ωραίο τρόπο, με εύκολο τρόπο και επειδή ακριβώς πρότεινα αυτές τις νέες προτάσεις για όνομα και είδα τις αντιδράσεις, θεωρώ ότι θα πρέπει μάλλον να επιλέξουμε την πρόταση αυτή δηλαδή γενιά για την Ευρώπη. Μία πρόταση η οποία νομίζω θα βρει μεγάλη υποστήριξη από όλους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αλή. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και την κυρία εισηγήτρια Νομίζω ότι η Επιτροπή μας πρέπει να τονίσει ιδιαίτερα το ότι ο έρασμος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απειλείται από περικοπές του προϋπολογισμού του. Να δείξουμε δηλαδή ότι δεν δεχόμαστε να θέσουμε σε κίνδυνο το πρόγραμμα αυτό. Ο έρασμος για όλους παίρνει νέα διάσταση σήμερα. Είναι πρόγραμμα που αφορά όλους τους Ευρωπαίους αλλά και παραπέρα. Και η δυνατότητα αυτή για όλους και όλες να μπορέσουν να εκπαιδευτούν σε χώρα άλλη από τη δική τους, όπως μας είπε και η Κομισιόν, σημαίνει ότι συμφιλιώνουμε τον κόσμο με την ιδέα της Ευρώπης. Σήμερα βλέπουμε ότι η Ευρώπη αφιερώνει μόνο 1% του προπλογισμού της για αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τι θα γίνει αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι. Αναρωτιόμαστε σήμερα μήπως δεν θα έπρεπε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός αυτός και επιμένω ιδιαίτερα για τους φοιτητές και φοιτήτριες που προέρχονται από πτωχές οικογένειες, διότι γενικά ο έρασμος πολλές φορές συχνά αφορά μόνον ελίτ που βγαίνουν από τις μεγάλες σχολές ή τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εγώ θα ήθελα το μήνυμα που θα δώσουμε να είναι σαφές ως προς τον προϋπολογισμό. Να πούμε δηλαδή ότι θέλουμε τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν αύξηση του προϋπολογισμού του Εράσμου. Σας ευχαριστώ άλλος κανείς εδώ μπροστά. Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η Καρή Μαντέλη για την διατήρηση του προϋπολογισμού του Εράσμου για όλους. Ιδιαίτερα σε μια στιγμή όπου η κατάσταση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, του ενωσιακού προϋπολογισμού απειλεί τον έρασμο γενικότερα γιατί δεν έχουμε κονδύλια για αυτόν πλέον. Επομένως όλα αυτά παίρνουν ιδιαίτερη αξία σήμερα και προσθέτω ότι πρέπει το πρόγραμμα αυτό να αφορά όλους τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα τους μαθητευόμενους για να μπορέσουν να υποφεληθούν όλοι από αυτήν την αυξημένη διεθνή ενωσιακή κινητικότητα γιατί είναι θέμα μέλλοντος της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Θέλω να προσθέσω κάτι. Καταρχήν ότι φυσικά ευχαριστώ την εισηγήτρια που επιτρέπει στην Επιτροπή μας να εγκρίνει μια ωραία γνωμοδότηση. Έπειτα αυτά από τα οποία είπε ο κύριος Μπακ, δύο σχόλια. Ένα, η συγχύτρια δεν προτείνει αλλαγή. Ξέρω ότι στην Επιτροπή Πολιτιστικών πολυσυζητιέται το θέμα. Συνεννοηθείτε με εκείνη. Δεύτερον όμως, εγώ διαφωνώ. Θα σας πω γιατί. Τα έχω ξαναπεί με την κυρία Μπλίνκ Τσιούτε και το απόγευμα. Αυτή τη φορά συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν για τον έρασμο για όλους. Μου λένε ότι αφορά τους φοιτητές ε, που έχουν κάνει δύο χρόνια σπουδών. Δεν είναι αλήθεια αυτό θυμάμαι από την προηγούμενη θητεία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι είχε διατυπωθεί μια πρόταση του Εράσμου για μαθητεία διότι ο Έρασμος λέγαμε είναι success story και εκεί βασίζεται η πρόταση της Κομισιόν. Μένα μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Ξέρω ότι η κυρία Δωρής Πακ δεν συμφωνεί Λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά δεν βρισκόμαστε σε περίοδο όπου επιτρέπονται όλα τα συντηρητικά προγράμματα. Κάποτε είχαν επιτυχία, αλλά πρέπει τώρα να ανοίξουν τα πράγματα, γιατί ζούμε σε μια περίοδο όπου το κύριο θέμα είναι να βοηθήσουμε τους νέους, να τους επιτρέψουμε να οργανώσουν κάποιο μέλλον και ο έρασμος είναι ακριβώς αυτό με βάση την πρόταση της Κομισιόν. Γι' αυτό υποστηρίζω πολύ στεναρά την εισηγήτρια να μην αλλάξει ο τίτλος, ακόμη κι αν υπάρξουν μερικές τροπολογίες που θα εγκριθούν, τέλο πάντων. Αυτά ήθελα να σας πω. Όπως λέω άλλωστε συνήθως όποτε αναφερόμαστε στην έκθεση της κυρίας Μπλικιβιτσούιτ, στην οποία ξαναδίνω το λόγο για να καταλήξει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής που τοποθετήθηκαν. Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς συζητήσαμε τις συνδεστικές προτάσεις από κοινού με μέλη και άλλων επιτροπών ε, και αποφασίσαμε ότι η πρόσβαση στο πρόγραμμα και στην κινητικότητα στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τονίζεται παρκώς τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει. Δηλαδή θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να είναι προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν τα επαρκή μέσα. Μια άλλη συμβιβαστική πρόταση αφορούσε τον προπολογισμό. Συζητήσαμε ιδιαίτερα το θέμα αυτό και έχουμε μια διάταξη βάσει της οποίας η χρηματοδότηση δεν μπορεί να είναι κατώτερη της σημερινής. Γιατί εδώ μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης. Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να μειωθεί. Και η χρηματοδότηση για ορισμένες ομάδες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτό που προβλέπετε αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020. Τώρα, σε ό,τι φορά την ονομασία. Είπα ότι δεν πρόκειται να προτείνω αλλαγή της ονομασίας, του τίτλου, του προγράμματος. Αυτό πρέπει να το συζητήσει η Επιτροπή Πολιτισμού και ο κύριος Κάστλερ και θα το συζητήσουμε αυτό με την Επιτροπή εκείνη. Εγώ πιστεύω ότι στο περιεχόμενο εκφράζονται οι κυρίες ιδέες ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει λοιπόν να είναι προσβάσιμο στους νέους αλλά και στις υπόλοιπες γενιές καθώς αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία και το βλέπουμε αυτό στην πράξη ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο δηλαδή το πρόγραμμα και πρέπει να το συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε το σύνολο των ε, τροπολογιών αύριο και η Επιτροπή Πολιτισμού θα αποφανθεί στις 6 Νοεμβρίου. Τώρα, φτάνουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, το σημείο 10. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ροντσούλη για την παρουσίαση των 17 ε, συμβιβαστικών τροπολογιών. Το σχέδιο γνωμοδότησης ε, είναι για την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Μπερνάντε την Βερνιόν εισηγήτρια. τροπής οδηγίας οδηγίε για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρηση για την εσωτερική αγορά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Σιλίκο. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφοι, το κείμενο που θα ψηφίσουμε αύριο αποτελεί ένα νέο βήμα προς ε, τον εξυγχρονισμό της ενιαίας αγοράς. Η αναθεώρηση της οδηγίας θα επιτρέψει σε πολλούς ε, επαγγελματίες να μπορούν να δραστηριοποιούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος, προσφέροντας ε, καλύτερες υπηρεσίες σε πάνω από 550 εκατομμύρια πολίτες μία επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας, μείωση του κόστους και ε, εις βάθος ε, γλωσσικός έλεγχος είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την νομοθετική πρόταση. Η εισαγωγή μιας ε, ευρωπαϊκής κάρτας αποτελεί ένα νέο μέσο για να ε, βοηθήσει την κινητικότητα των εργαζομένων ε, χάρη στη συνεργασία και τη διαθεσιμότητα όλων των συναδέλφων ήταν δυνατόν να καταλήξουμε στη σύνταξη 17 συμβιβαστικών τροπολογιών που ενισχύουν το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ για να έχουμε μεγαλύτερη κινητικότητα για τους εργαζομένους, καλύτερους ελέγχους και σβάθος και να προσδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των καταναλωτών. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, ε, οι συμβαστικές προτάσεις Α και L ε, επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να αρνηθούν όταν υπάρχουν κάποιοι λόγοι όπως υγεία των στενών κτλ. Στο σημείο Κ προτείνεται διαβούλευση των ε, κοινωνικών εταίρων ε, στην περίπτωση που υπάρχει έγκριση για αυτή την μερική πρόσβαση σύμφωνα με όσο ε, υποστήριξαν από τη μέλη και ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Συμβασμό Β αποκλεί του συμβολογράφου από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Ε, τώρα οι συμβαστικέ προτάσει Τ και Ο ενισχύουν αυτό που ζήτησε αυτή η Επιτροπή για να μπορεί ένας επαγγελματίας ε, να δραστηριοποιείται σε ένα άλλο κράτος μέλος, όμως είναι απαραίτητη η έλεγχη, δεν πρέπει όμως να εισάγουν διακρίσεις ή αρμόδιες εθνικές αρχές ε, οι κοινωνικοί εταίροι και οι διάφορες ενώσεις συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού των ελέγχων αυτών και ο συμβασμό D, ΔΕΛΤΑ, διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στην περίπτωση όπου ένα επαγγελματία εφίσταται πειθαρχικά μέτρα ή έχει εμ, καταδικαστεί και έχει αποκλειστεί, του έχει αποκλειστεί δυνατότητα να ασκήσει τα επαγγελματικά του καθήκοντα και προσωρινά και στου συμβασμού ε, G και P προβλέπεται μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων των εμπειρογνωμόνων, ε, των ειδικών στην προετοιμασία πιλωτικών σχεδίων και κατεξουδότηση πράξεων. Ο Συμβασμό F επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει κριτήρια ε, για την έκδοση αυτής της επαγγελματικής κάρτας ε, και ζητά μελέτη αντικτύπου και οι συμβέσεις H, I, G και A περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ε, σε αυτή την κάρτα. Αναφέρεται η προθεσμία των τεσσάρων ε, εβδομάδων στο ΕΜ προτείνεται συνεχής σύστημα κατάρτισης ε, για όλους τους εργαζομένους, για όλα τα επαγγέλματα και ο πιο αμφίσιμη συμβιβαστική τροπολογία, το Q, προτείνει μια μεταβατική περίοδο 6 ετών όπου τα κράτη-μέλη καλούνται να θετήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης για τις νοσοκόμε που θα ισούται με τα 12 έτη. Σας ε, ευχαριστώ όλους και αν ε, υπάρχουν συνάδελφοι που δεν συμφωνούν θα ξαναζητήσω το λόγο στο τέλος. Ευχαριστώ. Τέσσερις ακόμη έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν ναι, Ευχαριστώ Πρόεδρε και την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία και τις συμβιβαστικές τροπολογίες που επιτρέπουν μια καλύτερη εξισορρόπηση για το θέμα της κυκλοφορίας των εργαζομένων και τη δυνατότητα των χωρών μελών να μπορούν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. τα μέτρα που προτείνει επιτρέπουν καλύτερη διευθέτηση της, της διαμεθοριακής κινητικότητας. Να μπορεί κανείς δηλαδή να λάβει μια επαγγελματική μετεπέδευση και σε τη χώρα, σε χώρα άλλη από τη δική του. Επίσης προβλέπονται εγγυήσεις για εξαιρέσεις με βάση τον ορισμό των υπηρεσιών από τη σχετική οδηγία. Πρέπει να μπορούν οι Ευρωπαίοι να έχουν συνεργάτες που να μιλούν την ίδια γλώσσα με κίνους. Επίσης υπάρχει το θέμα της πληροφόρησης για το επαγγελματικό δελτίο ή κάρτα που επιτρέπει την καλύτερη διευθέτηση των κοινωνικών ε, διαμαχών στον τόπο εργασίας και την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων παντού. Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Η Νάντια Χίρς και μετά ο Θωμάς Μάν. Zusammenarbeit. Ich glaube, dass insgesamt ein Ευχαριστώ πολύ. Ήταν εξαιρετική συνεργασία και το αποτέλεσμα μου φαίνεται πολύ επικοδομητικό και πλούσιο. Όσον αφορά την τροπολογία J, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Η επαγγελματική κάρτα εδώ έχω την εντύπωση ότι συγκεντρώνονται πολλές πληροφορίες και θα υπάρξει και θέμα προστασίας των δεδομένων. Θα πρέπει να είμαστε πιο επιλεκτικοί και να σκεφτούμε ποια από αυτά τα στοιχεία ε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την κάρτα. Επίσης, όσον αφορά την συμβαστική πρόταση Q, Νομίζω ότι μπορέσαμε με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε ότι αν υπάρχει επαγγελματική κατάρτιση αυτή να συμπεριληφθεί, να ληφθεί υπόψη. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς κάποιος έφτασε σε μία κατάρτιση, πώς συγκέντρωσε κάποιες δεξιότητες, κάποια προσόντα και όχι ποια θα είναι αυτά. Όσον αφορά τη συμβαστική τροπολογία, που αφορά αυτή που υποβάλαμε με τον κύριο Τούρουνεν και αφορά τις μαθητίες, θέλουμε οι μαθητίες να αναγνωρίζονται. Και γι' αυτό και αυτό θα θέλαμε εδώ να συμπληρωθεί το κείμενο αυτό με την πρόταση ότι θα πρέπει να πληρώνονται. Δηλαδή, εδώ βλέπετε ότι κάποιος ο οποίος έχει κάνει μία ε, μαθητεία χωρίς μισθό, χωρίς καμία αμοιβή, δεν υπολογίζεται. Δηλαδή, έχει διπλό μειονέκτημα και έχει κάνει μία δωρεάν ε, μαθητεία και δεν του υπολογίζεται. Εδώ αυτό θα πρέπει να ε, διορθωθεί. Το Μασμάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνεργασία. Κάποια μπορώ να τα δεχτώ. Προσπαθούμε να αυξήσουμε την κινητικότητα. Τώρα, στην πράξη τι γίνεται. Βλέπουμε ότι εδώ προτείνονται διάφορες διάρκειες 10 χρόνια, 12 χρόνια. Τελικά βλέπετε όμως ότι κάποιος με ένα πτυχίο μετά από 10 χρόνια σχολείο θα πρέπει να δούμε τι προσόντα, τι δεξιότητες, τι mm. πραγματικές γνώσεις έχει. Εδώ προτείνεται να περάσουμε από 10 σε 12 χρόνια. Το θέμα είναι βέβαια να μην φτάσουμε σε μια μόνο ακαδημαϊκή αντιμετώπιση αυτών των ε, προσόντων και αυτοί οι οποίοι δεν βγαίνουν από το παραδοσιακό σχολικό σύστημα να μην λαμβάνονται υπόψη. Και στη Γερμανία έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ ποιοτικό θα έλεγα και το οποίο δεν βασίζεται καθαρά και μόνο σε ακαδημαϊκές γνώσεις. Χαίρομαι που στην Ισπανία ε, σας ενδιαφέρει αυτό το σύστημα. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να περάσουμε από τα 10 στα 12 χρόνια, σίγουρα. Και η τροπολογία που είχα υποβάλει 36 έγινε δεκτή, την έχει συμπεριλάβει. Νομίζω ότι εδώ σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό το ελάχιστο επίπεδο και εδώ θα αναφερθώ και στην τροπολογία 134 και 135. Η συμβαστική τροπολογία Q μου δημιουργεί όμως ακόμα πρόβλημα. Γιατί ποιος είναι ο σκοπός να περάσουμε από τα 10 στα 12 χρόνια. Αυτός είναι όμως ο σωστός τρόπος να γίνει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να τη δεχτώ αυτή την τροπολογία, τη συμβαστική Q. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Καλύτερη κατάρτιση. Να μην υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Δηλαδή να μην υπάρχουν δύο κατηγορίες και θα πρέπει σε όλα τα κρατημέλη να δίνονται αυτές οι δυνατότητες μετεξέλιξης και κατάρτισης. Ξέρω ότι τα προβλήματα δεν θα προκύψουν μόνο από τη Γερμανία. Σίγουρα και από το Λουξεμβούργο, από την Αυστρία, από την Ολλανδία. Τα βλέπουν τα πράγματα όπως και εμείς. Και σίγουρα αύριο αυτό θα φανεί. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να πλησιάσουμε η μεν τους δε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αυριανή πρόταση. Θα πρέπει να τελειώσουμε με τους ομιλητές. Η κυρία Σίμπελ, Άρκιν, Σλοβιέσκα και Χέντελ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Η Μπίργκιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις, όχι μόνο στην εισηγήτρια, αλλά και στην Επιτροπή, αν υπάρχει κάποιος παρόν. Όσον αφορά το θέμα της ε, συζήτησης στη Γερμανία, όσον αφορά την κατάρτιση, ναι, θα πρέπει να προσφέρονται δυνατότητες κατάρτισης, όπως αυτές που έχουμε στη χώρα μας, για τις οποίες είμαστε περήφανοι. Στη Γερμανία Υπάρχουν αυτοί που είναι κατά αυτής της υποχρέωσης για 12 ετή ε, κατάρτιση, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι υπέρ. Αυτοί δηλαδή που βρίσκονται σε αυτούς τους τομείς και σε αυτά τα επαγγέλματα είναι υπέρ του να ανυψωθεί το επίπεδο. Να υπάρχει δηλαδή 12 ετής ε, εκπαίδευση πριν φτάσει κανείς στην τριετή κατάρτιση. Και αυτό δεν σημαίνει αποκλειστικά και μόνο ένα ε, απολυτήριο λυκείου ή ένα μπακαλωρεά ή ένα αμπιτούρ. Το θέμα τώρα των γλωσσικών υποχρεωτικών απαιτήσεων. Ναι, παραδείγματο χάρη για μια νοσηλεύτρια είναι σημαντικό να μπορεί να συνεννοηθεί με τους ασθενείς. Το θέμα όμως είναι γιατί παραδείγματο χάρη για τους νοσηλευτές ζητάμε 12 ετή εκπαίδευση, στα άτομα όμως που παρέχουν ε, φροντίδα στους ηλικιωμένους, εκεί λέμε 10. Ξέρετε ότι χρειάζονται πολλές ε, δεξιότητες και προσόντα για αυτήν την κατηγορία εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λιγάκι πιο λογικοί στις προτάσεις μας. η κυρία Χάρκιν. Πρόεδρε, σύντομη θα είμαι γιατί δεν έχουμε χρόνο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική συνεργασία. Χαίρομαι πάρα πολύ με τον τελικό συμβασμό Α σχετικά με την μερική πρόσβαση για του επαγγελματίε στον τομέα τη υγεία. Νομίζω ότι βρίσκει μια καλή ισορροπία και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε. Επίσης, ε, Χαίρομαι που υθετήσετε τη δική μου διατύπωση σε σχέση με το αν ε, ένα ε, επαγγελματή δεν μπορεί να ασκήσει πλέον τι επαγγελματικέ του υποχρεώσει. Ε, χαίρομαι που έχετε συμπεριλάβει και τι προσωρινέ απαγορεύσει τι επαγγελματικέ και επίση χαίρομαι που δεχτήκατε τι περισσότερε τροπολογίε μου, αλλά για το συμβασμό J έχω μια ένα σχόλιο, θα συμφωνήσω με την συνάδελφο Νάντια μεταξύ των πληροφοριών που απαιτούνται για τις ε, κάρτες. Ε, νομίζω ότι εκεί έχουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες ε, και εκεί δημιουργούνται κάποια στήματα. Αλλά κατά τα λοιπά σας ευχαριστώ, είμαι ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Η κυρία Ιστοβλέσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη αναφέρθηκε το επιμέχο ζήτημα ε, για την περίοδο των 12 ετών. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά τι είπε ο κ. Μάν. Γιατί είναι κατά της δυνατότητας προσαρμογής ε, κατά τη διάρκεια μιας εξέτους περίοδου, γιατί αυτό προτάθηκε από την συγκήτρια στο συμβασμό Q. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε τον ε, κοινό παρονομαστή που δεν θα πρέπει να είναι ο κατώτερος αλλά ο ανώτερος. Νομίζω ότι η Γερμανία μας δίνει το καλό παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, ε, γιατί εσύ το μας διαφωνείς. Πραγματικά αυτό με προβληματίζει. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα επιλύεται με την περίοδο των 6 Γιατί δεν θέλει να πάει στα 12 έτη, νομίζω είπε, λέει η Πρόεδρος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. δεν θέλει το αποτέλεσμα, επομένως δεν θέλει καθόλου να μπει σε αυτό το δρόμο. Παρακαλώ. Ich kann jetzt nicht für Thomas Mann... Δεν θα μιλήσω εξ ονόματος του Τόμας Μαν, αλλά τα ίδια περίπου θα πω. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι 10 ή 12 χρόνια και αν θα έχει κανείς ένα πολιτήριο λυκείου, ένα αμπιτούρι, όχι. Αν κατάλαβα καλά, Πρόκειται για διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικά συστήματα. Κατάλαβα, μιλώντας μεγάλους συναδέλφους, ότι τα τελευταία δύο χρόνια αυτής της ε, δωδεκαετούς ε, εκπαίδευσης μπορεί κάποιος να επιλέξει κάποια μαθήματα και να εξειδικευθεί. Με μία επαγγελματική κατάρτιση, λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε κάτι αντίστοιχο. Κάτι που να γίνεται τα τελευταία χρόνια. Και μέχρι τώρα δεν γινόταν. Στην Ευρώπη έχουμε τελείως διαφορετικά συστήματα. Ναι. Δεν μπορεί όμως κανείς να πει ότι τα πράγματα είναι χειρότερα στη Γερμανία με 10 χρόνια υποχρεωτική κατάρτιση και σε άλλα ε, κράτη είναι καλύτερα με 12. Τι να σας πω, θα πρέπει εδώ να προσπαθήσουμε να πείσουμε οι μεν τους ναι και μιλάει για μια ευρωπαϊκή οδηγία. Αν περάσει το... η διάρκεια της εκπαίδευσης από 10 χρόνια σε 12, Αυτό θα πρέπει προηγουμένως να μας οδηγήσει σε μια σύγκριση των συστημάτων που είναι διαφορετικά διαρθρωμένα σε εθνικό επίπεδο και έχουν διαφορετικούς ε, σκοπούς. Βλέπετε ότι μια δωδεκαετής γενική ε, εκπαίδευση χωρίς καμία εξειδίκευση. Ναι, γιατί όχι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει προηγουμένως να δούμε το περιεχόμενο και τα ευρωπαϊκά πρότυπα που περιέχει αυτό, αυτή η 12 εκπαίδευση. Τώρα, όσον αφορά τη συμβαστική πρόταση Q, και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω. Μάλιστα. Έχουμε καθυστερήσει. Θα είμαι πιο αυστηρή. Θέλετε να παρέμβετε κύριε Δεσιλέρ. Ε, ωραία, δεν θέλετε. Πολύ ωραία. Για το συγκεκριμένο, όχι για... και για το μέλλον, κυρία Συγητρία. Θέλετε να εξαγάγετε κάποια συμπεράσματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σύγχυση και ίσως να προσεφηνήσω. Αναφέρουμε στον Τόμος ε, η τροπολογία σου υπαριθμών 36. Εγώ δεν σκοπεύω να την υποστηρίξω, γιατί ουσιαστικά έρχεται σε αντίθεση με όλη τη δουλειά που έγινε μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων για να φτάσουμε στο συμβασμό Q. Και έρχεται σε αντίθεση με όλο το έργο που μόλις σας εξέθεσα. Εγώ ήξερα ότι τελικά όλη η δουλειά που είχε, παρόλη τη δουλειά που είχε γίνει για το συμβασμό Q, ε, θα κινδυνεύαμε να χάσουμε και τα θετικά και θα καταστρέφαμε τη δουλειά μηνών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συμβασμό Q, το είπα με βλέπετε εδώ, εκφράζομαι με ιδιαίτερο πάθος γιατί πριν να γίνω βουλευτής, εγώ ήμουν ε, επικεφαλής όλου του προσωπικού που απασχολείται στον ε, τομέα της υγείας σε ένα μεγάλο νοσοκομείο στην Ιταλία. Ξέρω λοιπόν τι σημαίνει η κατάρτιση των νοσηλευτών και δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια η νοοτροπία του να θεωρούμε αυτό το επάγγελμα, να βλέπουμε αυτό το επάγγελμα να θεωρείτε ότι απλώς ε, είναι ένας τρόπος να φτάσει κάποιος να αποκτήσει μια θέση εργασίας. Αυτό με υπογοητεύει. Κοιτάξτε, το να είναι κάποιος επαγγελματίας νοσοκόμος ε, είναι αποστολή. Δεν είναι ένας τρόπος να βρει απλώς κάποιος μια δουλειά γιατί έχουμε έλλειψη σε νοσοκόμους. Έτσι λοιπόν, ε, δεν μπορούμε να μειώνουμε ή να αυξάνουμε το επίπεδο της κατάρτισης για να λύσουμε το θέμα της απασχόλησης. Εγώ νομίζω ότι όλοι εμείς εδώ θα πρέπει να κάνουμε, αν κάναμε μάλλον την ίδια συζήτηση για τους γιατρούς, κανένας από εσά και αναφέρουμε στους Γερμανούς συναδελφούς δεν θα ονειρευόταν ποτέ να ε, μειώσει τα έτη που για την εκπαίδευση των γιατρών. Το ίδιο ισχύει και για τους νοσοκόμους, γιατί αν ε, κάνουν λάθος, ποιος θα πληρώσει. Εδώ μιλάμε για τη ζωή του ασθενούς. Έτσι λοιπόν, αν ε, παρελόγω αύριο η Επιτροπή παρουσιάσει ένα κείμενο όπου θα λέγεται ότι επειδή υπάρχουν ε, λίγοι γιατροί, επειδή δεν υπάρχουν ε, πολλές θέσεις εργασίας, μειώνεται τα χρόνια της κατάρτισης για τους γιατρούς, θα γινόταν επανάσταση. Έτσι λοιπόν, αυτή η αρχή πρέπει να ισχύει και για τους νοσοκόμους. Και κοιτάξτε, αν τα κατάφερε η Ιταλία, μπορεί και η Γερμανία να τα καταφέρει να προσαρμοστεί. Και συμβιβασμό του που βλέπετε εδώ, την ε, συμπερίληψη των έξι ετών, είναι ο πιο λογικός συμβιβασμός. Γιατί σε έξι χρόνια δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της οικονομική κρίσης, αλλά έχετε έξι χρόνια για να μπορέσετε να προσαρμοστείτε σε αυτήν την οδηγία. Και για μένα ε, είναι ο μεγάλος συμβασμός που βρήκαμε αυτός. Σε ό,τι αφορά τώρα τους νοσοκομούς που απασχολούνται στα γυροκομεία. Δεν υπάρχει στη δική μου χώρα μια τέτοια διάκριση, απλά μιλάμε για ένα νοσοκόμενο νοσηλευτή για όλους. Έτσι λοιπόν, ίσως ε, αυτό το θέμα αφορά περισσότερο τις ε, χώρες όπου υπάρχει αυτή η διάκριση, ώστε μπορούσαμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη τροπολογία προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενίσχυση του ελέγχου των γλωσσικών γνώσεων ε, και μάλιστα στον τομέα της υγείας ενισχύθηκε και τροποποιήθηκε αυτό το κείμενο υπέρ ε, αυτού του επαγγέλματος που δεν είναι τόσο λεπτό. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Σα ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τελικά λοιπόν το θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων περιορίζεται σε ένα πρόβλημα. Πρέπει 10 ή 12 χρόνια να επιμορφώνονται οι νοσοκόμες. Αιρωνικά ε, το λέω, αλλά επί, επ' αυτού σημειώνονται οι περισσότερες διαφωνίες. Υπάρχουν όμως και μερικά άλλα θέματα και θα τα λάβει υπόψη η συγκήτρια. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε αύριο και φτάνουμε στο τελευταίο μας σημερινό σημείο. Το 12 η εξέταση των τροπολογιών για την εξέταση της έκθεσης Αρτιέ για την περίφημη πρόταση για την ασφάλεια και υγεία όσο αφορά την εκκρίση των εργαζομένων σε κινδύνου προερχόμενου από φυσικού παράγοντε παρένθεση ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ας μην επανέλθω σε ολόκληρο το ιστορικό του θέματος. θυμίζω απλώς, παρακαλώ όσο θέλει να φύγει να το κάνει ησύχω. Και στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Tak, tak, Είχαμε λοιπόν παρατείνει τη διορία κατάθεση τροπολογιών για να σεβαστούμε τη διαδικασία του Συμβουλίου και δίνω το λόγο τώρα στην εισηγήτρια για να μας παρουσιάσει γιατί υπάρχουν 249 τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξαναπιάνουμε λοιπόν αυτή τη δουλειά αφού το Συμβούλιο άλλαξε στάση με την αλλαγή των διαφόρων εναλλασσομένων προεδριών γιατί μερικές βασίστηκαν στο κείμενο, άλλες στις προσθήκες και έτσι δημιουργήθηκαν πολλές δυσκολίες για μας γιατί οι διαδικασίες συνεχώς άλλαζαν κάθε έξι μήνες δηλαδή. Τέλος πάντων, 233 τροπολογίες κατατέθηκαν σε πρώτη φάση από τις πολιτικές ομάδες, ένα τρίτο από τους πράσινους. Μετά ξανάρχισε να τρέχει η διορία κατάθεσης τροπολογιών και σας ευχαριστώ γιατί τελικά μπόρεσα να επανυποβάλω 16 τροπολογίες συμπληρωματικές ώστε με βάση όλη την εργασία που είχαμε κάνει στην ομάδα εργασίας του Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί δηλαδή τις θέσεις όλων των βουλευτών να καταλήξουμε σε κάποια σύγκληση. Οι τροπολογίες αυτές αφορούν πρώτον την απαραίτητη εξισορρόπηση μεταξύ προστασίας των εργαζομένων και της πιθανής χρησιμοποίησής τους στον ιατρικό τομέα. Πολλές τροπολογίες από όλες τις πολιτικές ομάδες γι' αυτό μιλούν. Τη θέληση αυτή δηλαδή να διατηρηθεί και να ενισχυθεί θα έλεγα η προστασία των εργαζομένων που υφίστανται ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Και απ' την άλλη, η οδηγία αυτή του 2004 ποτέ δεν μπόρεσε να εμφαρμοστεί και θελήσαμε να δούμε γιατί. Κάτι άλλο που για το οποίο μιλούν πολλές τροπολογίες αφορά τις συνταγές ή τα ελάχιστα όρια. χωρίς να υπάρξει η παναχώρηση, τα ελάχιστα όρια, η παναχώρηση στα ισχύοντα. Αυτός είναι δεύτερος μεγάλος άξονας των τροπολογιών. Τρίτος, κάτι δύσκολο, η θέλησή μας να λάβουμε υπόψη μας τις συνεχείς τεχνικές προόδους που σημειώνονται στη χρήση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και απ' την άλλη τους περιορισμούς που έχουμε όλο και περισσότερο στην, που μας επιβάλλονται για θέματα τεχνολογικών προόδων. Άλλος άξονας των τροπολογιών είναι η χρήση προσθετικών στοιχείων στο σώμα που πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη αν υπάρχει μάλιστα έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Άλλος άξον, ο καθορισμός ορισμένων κατευθυντηρίων γραμμών για τη χρήση που υπάρχουν σε ορισμένες χώρες όπως την Ολλανδία όπου υπάρχουν οδηγίες χρήσεως που εξυπηρετούν πολύ τους αρχηγούς, τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τους υπεύθυνου γενικότερα για την προστασία του προσωπικού, οδηγίες χρήσεως που αφορούν και την ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο, την ασφάλεια δηλαδή των προσώπων και του προσωπικού. Έκτος άξον των τροπολογιών η πιθανή αναθεώρηση του κειμένου. Αν θα καθορίσουμε δηλαδή, αν θα το θεωρήσουμε βράχη πρόθεσμο ή αν προβλέψουμε ότι μπορεί να αναθεωρηθεί με βάση νέα στοιχεία, πρόοδο, έρευνα πρέπει και από αυτού να συμφωνήσουμε μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αυτός λοιπόν ήταν ο έκτος άξον και έβδομος οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στα, της έκθεσης ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Έτσι συνοψίζω τις κατηγορίες των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί από τις πολιτικές ομάδες. Προσθέτω δε τις 16 τροπολογίες που προστίθενται σε αυτές από μένα. Η τροπολογία 234 αφορά το σκεπτικό και μιλάει για την παραπομπή στην οδηγία για την εφαρμογή, της εξαίρεσης για την εφαρμογή της οδη, προηγούμενης οδηγίας 2004-144 και που καθορίζει στην 31η Δεκεμβρίου 13 το όριο της εξαίρεσης από την προηγούμενη οδηγία. Πρέπει λοιπόν πολύ πριν από τότε να έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Και σας υπενθυμίζω ότι θέλουμε εδώ να καταλήξουμε. Δεύτερη τροπολογία 235 από τις 16 Εδώ βάζω ένα στόχο για την ασφάλεια των εργαζομένων που υφιστανται ηλεκτρομαγνητικά πεδία και περνάμε στη 236 για το συγκεκριμένο τομέα των ενόπλων δυνάμεων. Να υπάρχουν ειδικά μέτρα προστασίας για τις ένοπλες δυνάμεις και την έκθεσή τους ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως από το ΝΑΤΟ. 237 για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων της έκθεσης τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση πάντα για την ασφάλεια των δεδομένων 238 εδώ αναφέρουμε τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και το ονομάζουμε safety risks. Μετά το επόμενο ιατρική κίνδυνη, κίνδυνη για την υγεία από τη χρησιμοποίηση διαφόρων προσθέσεων. Μετά, μετά λέω, ζητούμε διαβούλευση με ειδικό, θα ζητήσουμε την επόμενη πέμπτη συνεννόηση με τους διάφορους σκιώδεις από τις ομάδες για να δούμε τι τιμές πρέπει να βάλουμε και όρια που θα συμφωνήσουμε στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Μετά η επόμενη είναι απλοποίηση, το πεδίο εφαρμογής δηλαδή. Το 240 ζητάει ενδυνάμωση γιατί η οδηγία δεν μιλάει καθόλου για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά Το 241 ενδυναμώνει το ρόλο του εργοδότη και την ευθύνη του. Το ίδιο και το 242. Το ίδιο. 243 καθορίζει πώς θα, θα μεταφραστούν αυτά στον εθνική νομοθεσία και η 245 καθορίζει διάφορες εξαιρέσεις για το άρθρο 3 επί των οριακών τιμών έκθεσης. Η εξαίρεση για τις ιατρικές εξετάσεις ηλεκτρομαγνητικού πεδίου καθορίζεται περαιτέρω 247 στο 248 άλλες ειδικέ εξαιρέσεις και νομίζω ότι έτσι ε, τελείωσαν αυτές ήταν οι τελευταίες τροπολογίες ώστε την επόμενη φορά να μπορούμε, αφού έχουμε δει τον ειδικό την επόμενη πέμπτη, να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Ευχαριστούμε Σιλβάνα Ράπτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ωραία μας τα είπε η εισηγήτρια. Την ευχαριστούμε για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ε, πάμε πιο γρήγορα τώρα και αυτό είναι ένα καλό πράγμα, είναι μια καλή εξέλιξη. Ε, είδα και το ρολόι κυρία Πρόεδρε και ξέρω και είμαι σύντομη πριν μου το πείτε. Ε, λέω λοιπόν τα εξής από τις τελευταίες τροπολογίες που έχει καταθέσει η συγγήτριά μας. Ε, τις βρίσκουμε γενικά σε μια καλή κατεύθυνση. Ωστόσο υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει, στα οποία θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Μακροχρόνιες συνέπειες. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή επιστημονικά δεδομένα που να μας διαβεβαιώνουν ότι υπάρχουν μακροχρόνιες συνέπειες. Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν είμαστε και ήσυχοι ότι τίποτα δεν συμβαίνει. Και στο σημείο αυτό δίνω ένα παράδειγμα, το οποίο μάλιστα έχει σχέση και με ένα θέμα που θα συζητήσουμε αύριο. Μιλάω για τον αμίαντο. Για τον αμίαντο ποτέ δεν υπήρχαν μελέτες, ήμασταν όλοι ήσυχοι, χτίζαμε τα σπίτια μας, ε, χτίζαμε κτίρια, χτίσαμε το κτίριο εκεί της Κομισιόν το οποίο ήταν γεμάτο αμύαντο και ξαφνικά είδαμε ότι υπάρχουν συνέπειες. Επειδή δεν θέλουμε να συμβούν τέτοια πράγματα και εδώ, γι' αυτό το λόγο είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, να παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και να είμαστε πώς να το πω, να είμαστε alert ώστε να λάβουμε αμέσως δράση. Διότι να μην ξεχνάμε ότι ε, στο, στο, η, κεντρική ε, ιδέα της οδηγίας και της δουλειάς που κάνουμε συνολικά εδώ είναι η πρόληψη. Ε, με το ίδιο πνεύμα αντιμετωπίζω και τον, το, το, τις τροπολογίες και την όλη τοποθέτηση πάνω σε αυτό που λέμε γνωστές επιπτώσεις στην υγεία. Είναι το ίδιο πνεύμα με το οποίο το αντιμετωπίζω. Ένα άλλο θέμα είναι το ξεπέρασμα των ε, τιμών, των ορίων της έκθεσης σε ορισμένες, το λέω μέσα σε εισαγωγικά, ε, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο, όμως ε, έχω το ερώτημα και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε όλοι μαζί ε, ποιος θα ορίζει, ποιος θα καθορίζει τι είναι το δεόντος αιτιολογημένο. Ε, παρουσιάζω μερικές μόνο από τις ε, ανησυχίες, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, από τις ανησυχίες μας και ε, μερικές από τις ε, έγνοιες μας, τις μέρημνες που πρέπει να έχουμε ε, για τους πολίτες. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ε, ένα καλό, να, έρθουμε σε ένα καλό τέλος σε αυτή την υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό ότι πια έχουμε όλες τις τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικό ότι επιτέλους θα έχουμε τον expert, τον ειδικό που θα μπορέσει με τις απαντήσεις που θα μας δώσει να μας διαβεβαιώσει για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα και βεβαίως περιμένουμε τις συμβιβαστικές που θα κάνει η εισηγήτριά μας, να τις δούμε με όλη την καλή διάθεση για να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες είτε είναι εργαζόμενοι σε περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είτε είναι ασθενείς. Σας ευχαριστώ. Θα σας δώσω συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να σας ζητήσω να μην μακρηγορείτε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η κυρία Ντελή. Κάρι Ντελή. Σας ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια για την διαδικασία που ακολουθήθηκε και για τη συνεργασία μας. Ε, πολύ τη διαφάνεια από την αρχή και την ευχαριστώ πολύ. Εγώ μόλις ανακάλυψα τη θέση του Συμβουλίου που εκ πρώτης ε, όψεως ε, φαίνεται ισορροπημένο το κείμενο, όμως δεν έχω δει ακόμη το κείμενο λεπτομερώς, θα το πράξω βεβαίως και ελπίζω ότι θα μας δοθούν κάποιες διευκρινήσεις και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς. Επιμένω ότι είναι επιτακτική ανάγκη γιατί χάσαμε πάρα πολλούς μήνες για την έκθεση αυτή, για αυτή την οδηγία και δεν μπορούμε να περιμένουμε ακόμη μήνες. Ε, ας κάνουμε ε, κάποιους καλούς συμβασμούς, καταλήξουμε σε καλούς συμβασμούς, ας ακούσουμε τις εμπειρογνώμονες και σημειώσουμε πρόοδο. Κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ρεαλιστική της προσέγγιση και θα πρέπει να το συστήσουμε αυτό μέσα σε 12 μήνες και νομίζω ότι τώρα αρχίζουν να συγκλίνουν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε που συμφωνούμε και στο πλαίσιο αυτό ανυπομονώ να συναντηθώ και με τους εμπειρογνώμονες να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ένα τελικό σχόλιο. Σας ευχαριστώ για ορισμένες από τις τροπολογίες που παρουσιάσατε. Νομίζω ότι επιλύουν κάποια από τα ζητήματα που μας αφορούν ιδιαίτερα και όπως το θέμα της περέκκλησης για το MRA και για τα ηλεκτρομαγνητικά δηλαδή παιδεία και όχι μόνο για τους ε, ε ίδιους ε, τους εργαζομένους αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε και σε κάποια βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα τα οποία δεν το γνωρίζουμε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο θέματα και εκτιμώ και τα σχόλιά σας ε, για το θέμα της αναθεώρησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξέρω ότι ε, η σάρωση, το σκάνινγκ, ε, δεν είναι η μόνη πηγή ε, ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις είχα ρωτήσει, είναι δύο εμπειρογνώμονες μας είχαν προσφέρει τις συμβουλές τους αν τώρα θα ήταν ικανοποιημένοι με την πρόταση που έχει κατατεθεί. Και έτσι λοιπόν όταν επέστρεψα στην πατρίδα μου διαβουλεύτηκα με έναν εμπειρογνώμονα στην Αγγλία τον ε, Dr. Κλίβενεν, ο οποίο ε, ήταν σύμβουλος και μας είπε ότι αν τότε ε, περνούσε η πρόταση έτσι όπως είχε προταθεί, τότε ναι, αλλά από τότε έχουν υπάρξει αυτές οι νέες τροπολογίες και τώρα υπάρχουν προβλήματα. Θα παρουσιάσω τέσσερα. Τροπολογία πέντε θέτει το όριο της ε, ε, στην ε, ιατρική χρήση της, του MRI, αλλά και οι υπόλοιπε χρήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην παρέκκληση, έτσι ώστε τα σκάνερ να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και να ευνοήσουν τους πάντες στην Ευρώπη. Η τροπολογία 23, που φαίνεται είναι ίδια με την 76 και την 179 ε, σχολιάζει το προτινόμενο χρονικό διάστημα των πέντε ετών για την παρέκκληση. Όμως ε, δεν ε, υπάρχουν νέες, νέα αποδεικτικά στοιχεία μετά την εφαρμογή και αν υπάρχουν νέα αποδεικτικά στοιχεία η Κομισιόν πάντοτε έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την οδηγία και η τροπολογία 28 αναφέρεται στις στρατιωτικές χρήσεις ε, όμως υπάρχουν ήδη διεθνή πρότυπα για να διασφαλίσουν την προστασία των εργαζομένων από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Έτσι λοιπόν δεν φαίνεται να είναι σκόπιμη εδώ. Τώρα η τροπολογία 73 αναφέρεται στην πρόταση να υπάρχει ελάχιστη υπόσταση από την πηγή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων αλλά έτσι θα καθιστούσε το MRI αδύνατο καθώς η SARS αποτελεί την πηγή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Ε, ο περιορισμένος χρόνος της έκθεσης ε, δεν είναι σχετικός ε, καθώς είναι τα όρια της έκθεσης ε, δεν μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε ένα μέσο όρο. Αυτά είναι ορισμένα από τα σημεία από τον εμπειρογνώμονα στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Σοφοκλέου θέλετε να πάρετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ζητήθηκε από την Προεδρία του Συμβουλίου, όπως παρουσιάσει εν συντομία στην Επιτροπή σας σήμερα, τα αποτελέσματα του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο. On behalf of the Presidency of the Council, we would like first of all... Εξ ονόματος ε, της Προεδρίας του Συμβουλίου, καταρχήν σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας και θα θέλαμε να σας ε, παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης της 4 Οκτωβρίου. Οι Υπουργοί έλαβαν κάποιες αποφάσεις σε αυτό το πολύ περίπλοκο και τεχνικό θέμα. Από την αρχή της Προεδρίας της Κύπρου θέσαμε σαν προτεραιότητα να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η έγκαιρη έγκριση αυτής της πρότασης γίνεται εφικτή είναι λοιπόν μεγάλη πρόκληση αυτή η απόφαση του Συμβουλίου. Εργαστήκαμε σκληρά, με πίεση χρόνου σημαντική. Είμαστε όμως τεπισμένοι ε, ότι η απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας των Υπουργών είναι η καλύτερη συμβιβαστική πιθανή λύση. Καταρχήν, αναγνωρίζει το Συμβούλιο ότι η πρόταση αυτή είχε σαν σκοπό, κύριο σκοπό την προστασία των εργαζομένων και την ίδια ώρα αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίσει κανείς την εφαρμοσιμότητα αυτής της οδηγίας. Το κείμενο του Συμβουλίου βασίζεται στις αποφάσεις της Αρμόδιας Επιτροπής για τις Ακτινοβολίες και ακριβώς επειδή πρόκειται για την αρμόδια αρχή, για τις ηλεκτρομαγνητικές ε, ακτινοβολίες και παιδεία, έλαβε υπόψη της τις γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και όλες τις τεχνικές πλευρές αυτής της πρότασης. Πιστεύουμε ότι αυτή η εμπειρογνωμοσύνη υψηλού επίπεδου φαίνεται από το κείμενο. Το κείμενο του Συμβουλίου Δείχνει επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για κάποιες αποκλήσεις και εξαιρέσεις από τα όρια που έχουν τεθεί σε κάποιες ειδικέ ε, περιπτώσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας των εξοπλισμών ηλεκτρομαγνητικής ε, και βεβαίως θα πρέπει να συνεχιστούν οι δραστηριότητες στον τομέα αυτό κάτι που επιτρέπει ότι σε αυτές τις πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και με την απαραίτητη αιτιολόγηση μπορεί να ξεπεραστούν τα όρια και να δοθούν κάποιες εξαιρέσεις την ίδια ώρα σε κάποιες περιοχές και για την χρήση των ενόπλων δυνάμεων μπορεί να δοθεί άδεια για τη χρήση αντίστοιχου εξοπλισμού. Οι εργαζόμενοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προστατεύονται από αρνητικές ε, συνέπειες. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η γενική προσέγγιση της απόφασης ε, του Συμβουλίου της προηγούμενης εβδομάδας είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος, ένα σημαντικό βήμα για να βρεθεί μια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια ποιοτική απόφαση, κάτι το οποίο δείχνει την ισορροπημένη προσέγγιση μας και τη λήψη υπόψη των ε, προτάσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ε, συμφωνία σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας τους επόμενες μήνες. Ναι, πίεση χρόνου. Έχετε ε, δίκιο, οι διερμηνείς μας έδωσαν πέντε λεπτά. Κυρία Σαρκή, έχετε μόνο δύο λεπτά να ολοκληρώσετε. Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν, Πιστεύω ότι όντως ε, έγινε ένα σημαντικό βήμα με την απόφαση της 4ης Οκτωβρίου του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι όλοι οι σκιώδεις εισηγητές επιθυμούν να κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτό το αδιέξοδο που υπάρχει από το 2004. Θα είμαστε όλοι περήφανοι για μια τέτοια απόφαση και σας ευχαριστώ πολύ όλους. Alors, Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Στις 19 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε τυχόν συμβιβαστικές τροπολογίες. Τελειώσαμε σήμερα με τις εργασίες μας και θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί σε 9.